Good morning. morning everybody. Good morning. Morgen. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Περιμένουμε προσέλευση μεγάλη σήμερα ή να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, η ημερήσια διάταξη την έχετε λάβει. Θέλω να σας γνωστοποιήσω τις εξής αλλαγές. Η συνεδρίαση των συντονιστών θα γίνει σήμερα 3 με 4 το απόγευμα και όχι το βράδυ. Παρακαλώ να είστε παρόντες. Χρειάστηκε να το κάνουμε αυτό λόγω ενός αιτήματο ε, συγκεκριμένου ε, συναδέλφου που αλλιώς δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στην σημερινή μας συνεδρίαση. Λοιπόν, το σημείο 16 θα το δούμε στις 3, το 9 στις 5 ε, και 4 και το 10 στις 5 ε, και 45. Γλώσσες είναι οι γνωστές, μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδριασή μας και περνάμε στο σημείο 3. Κατάσταση στην Ουγγαρία. Έχουμε να ψηφίσουμε μία γνωμοδότηση που συνέταξα εγώ για μια έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχω τοποθετηθεί, τα έχουμε συζητήσει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία λοιπόν. Έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας σας μαζί σας. Παρακαλώ βάλτε τις στις συσκευές σας. Αποσύρθηκαν ε, δύο τροπολογίες, η 8 και η 49. Και ξεκινάμε με την τροπολογία 23 υπέρ, κατά. Ψηφοφορία κάνουμε, ε. υπέρ, κατά, αποχές, όχι. Ας πάμε να ψηφίσουμε κατευθείαν ηλεκτρονικά για να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, μπορούμε να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίστε επί της τροπολογίας 26. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας είμαστε βέβαιοι καλύτερα. Πράγματι εγκρίνεται. Άρα 8 υπέρ, 8 κατά, άρα απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, Κατά. Μάλιστα. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Επί της τροπολογίας 35. 35. Πέρας. Απορρίφθηκε. Μεγάλη διαφορά. 36 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Απεσύρθη, όχι. Υπέρ, κατά, αποχές. Καλύτερα να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 4 απεσύρθη. Όχι, συγγνώμη, δεν απεσύρθη. Υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8-9 απεσύρθηκαν. 10 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά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 12 υπέρ, δύο εποχές. Ευχαριστώ πολύ. Α, ναι, υπερψηφίζει και ο συνάδελφος Τσέλερ, χωρίς την κάρτα του. Ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Χρειαζόμαστε τον συνάδελφο Βόρν θα ήταν καλό να ήταν παρόν. Μπορεί να μας ενημερώσει η πολιτική ομάδα των σοσιαλιστών πότε μπορούμε να περιμένουμε τον κύριο Βόρν. Είναι καθοδόν, μάλιστα, ωραία. Εντάξει, περνάμε στο σημείο 5 τότε. Επίσης δεν είναι εδώ η συγγήτρια. Ε, δεν μπορώ να ξανακάνω ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση για την Ουγγαρία. Τι να κάνουμε. Ε, συνάδελφε Πυρίνσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, κατάλαβα καλά, μιλάμε για, συζητάμε το σημείο 5. Το πρόβλημα είναι ότι η συγκίτρια είναι η Ίνες και δεν είναι ακόμα παρούσα. Α, μου ζήτησε, λέει ο κ. Πυρίνσκι, ελεγκτικό συνέδριο Παιδιά, 9 η ώρα αρχίζουμε. Ξέρετε ποτέ είναι 9. Όταν γράφει εκεί 9 και δίπλα 2 μηδενικά, αυτό είναι 9 η ώρα το πρωί. Und zwar υπήρχε ένας βουλευτής που έκανε μεγάλη φασαρία όταν καθυστερούσαμε πέντε λεπτά να αρχίσουμε τη συνεδρίαση και υπολόγιζε πόσο μας κοστίζουν οι διερμηνείς που έχουν βάλει το κοντέρ και μετράει από τις 9. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να τα ακούν αυτά και τα μέλη της αντιπροσωπείας. Τι να κάνω τώρα. Πρέπει να είναι εδώ οι παρόντες οι αρμόδιοι. Ποιος νομίζει ότι κάνω τη συνεδριάση για μένα. Ε, λάθος είναι αυτό. Ja gut, also ähm, genau. Der Kollege Vaughn, wann, wann kommt er denn? Ο κύριος Βόν, έχετε καμία ιδέα τι ώρα θα έρθει? Auto. Mm -hmm. Α, είναι καθοδόν. Καλά. Στα διάφορα έχετε τίποτα κανένα διάφορο να πούμε μέχρι να έρθουνε. Ούτε στα διάφορα δεν έχουμε. Η διοίκηση να το σκεφτεί. Μήπω ε, θα είχε νόημα να χαρίσαμε από ένα ρολόι σε κάθε βουλευτή. Τι να κάνουμε τώρα. Με πόνο καρδιάς πέντε λεπτά διάλειμμα. Περιμένουμε να καταφτάσουν οι αρμόδιοι. Ενδεχομένως στο ελεγκτικό συνέδριο, ο συνάδελφος Βον Ja, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Κατέφτασε όμως ο συνάδελφος. Επομένως, μπορούμε να δούμε το θέμα για την επιστολή στην Αλβανία. Η αρχική Αρχικά είχε σχεδιαστεί να πάμε και στη Φύρομ, όμως εγκαταλείφθηκε αυτό το σχέδιο. Κύριε Βόν, έχετε το λόγο να μας παρουσιάσετε την αποστολή στην Αλβανία. Ζητώ συγγνώμη, ήμουν ε, που ήρθα αργοπορημένος. Ε, ναι, <clears throat> αυτή η αποστολή στην ε, Αλβανία. Στην αρχή είχαμε πει να πάμε στην ε, ε, Αλφανία και στην με Παύλα, Μακεδονία ε, και ε, με μία φορά να κάνουμε τα πάντα. Ε, εν πάση περιπτώσει, εμείς είπαμε τελικά ότι δεν άξιζε τον κόπο και τελικά αποφασίσαμε να πάμε μονάχα στην Αλβανία. Έγκαιρη αυτή η επίσκεψη γιατί την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίστηκε η έναρξη των συνομιλιών για προσένταξη με την Αλβανία και βεβαίως ε, ε, σύμφωνα με την έκθεση ε, του 2016 του ελεκτικού Συνεδρίου υπάρχουν ακόμα ζητήματα τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να λυθούν. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις διαφθοράς. Αυτά όλα είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Πάντως το πρόγραμμα φαίνεται να είναι το να ήταν ε, καλό. Έχουν υποβληθεί πολλές ε, προτάσεις, επισκέψεις σε Υπουργεία, επισκέψεις ε, σε αρχές. Στριμώξαμε πολλές συνεδριάσεις και θα ήθελα να ε, παρακαλέσω τους συναδέλφους να κάνουν την προσπάθεια να έρθουν στην ε, ε, αντιπροσωπεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή αντιπροσωπεία, να έχουμε καλά ζητήματα και καλές θέσεις να συζητήσουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε κάποια μέλη τα οποία θα είναι παρόντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ και πολύ καιρό διαπιστώνουμε ότι η προθυμία των συναδέλφων να συμμετέχουν σε τέτοιες αποστολές δεν είναι και τεράστια. Καλωσορίζω τον κύριο Τσίγλερ, τμήματάρχη, αναπληρωτή τμήματάρχη για την Αλβανία, Βοσνία, ε, Ζεχοβίνη. Από τη Γενική Διεύθυνση ΝΙΑΡ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχετε μέσα λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλε. Χαίρομαι για την ευκαιρία που έχω να σας δώσω λίγο το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεών μας με την Αλβανία. Ήδη από το 2008 ε, είχαμε απελευθέρωση ε, διαβατηρίων. Το 2009 κατέθεσε αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2010 κάναμε τη γνωμοδότηση και είπαμε ότι για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις προενταξιακές ε, χρειάζονται 12 ε, προϋποθέσεις. Μετά από τέσσερα χρόνια το 2014 το Συμβούλιο ε, έδωσε ε, το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Είχαν απομείνει πέντε προτεραιότητες, οι επτά είχαν διεκπεριωθεί και το 2016 το Νοέμβριο με το προηγούμενο πακέτο διεύρυνσης υπό όρου το Συμβούλιο συνέστησε να αρχίσουν οι προενταξιακές διαπραγματεύσεις και οι όροι ήταν να υπάρχει αξιόπιστη και απτή πρόοδος στο διορισμό των δικαστών αυτό ε, κοιτάμε ε, ε, και θα το κοιτάξει και την προσωπία. Είναι το πρόγραμμα διορισμού και λειτουργίας του κασιστικού συστήματος και για πρώτη φορά υπάρχει παρακολούθηση διεθνής. Έχουμε έπτα δικαστές και εισαγγελείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν Αμερικανό. Ε, και θα μελετηθούν ε, οι ε, σχέσεις των δικαστών που είναι 800 στην Αλβανία και πλέον γιατί οι σχέσεις έχουν με το οργανωμένο έγκλημα, με τη διαφορά, αν έχουν επαγγελματική επάρκεια κτλ. Είναι έλεγχος γενικά της δικαιοσύνης. Έχουμε ήδη 20 δικαστές και εισαγγελείς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν από το δικαστικό σύστημα. Ορισμένοι απολύθηκαν από αυτό το όργανο, ε, ενώ άλλοι υπέβαλαν την παρέτησή τους για να μην υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο που είναι δημόσια διαδικασία και φέρνει πολλά πράγματα στο φως. Δηλαδή γίνεται τεράστια προσπάθεια κατά πολέμηση τη διαφθορά στην ίδια τη δικαιοσύνη. Ε, θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε με τους διεθνείς παρατηρητές. Έχει αρχίσει αυτή η προσπάθεια και πολύ ενδιαφέρον να το δείτε και συνδέεται πάρα πολύ και με το πολιτικό πρόγραμμα. Αυτή ήταν η προϋπόθεση, ο έλεγχος του δικαστικού συστήματος. Η Αλβανία έχει δώσει λοιπόν ε, τα αποτελέσματα που επιθυμούσαν και μόλις την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την πλήρη σύσταση ανεφόρων και προϋποθέσεων να αρχίσουν οι προενταξιακές διαπραγματεύσεις γιατί θεωρήθηκε ότι έχει πληρωθεί και αυτό το κριτήριο για τις υπόλοιπες πέντε, πέντε βασικές προτεραιότητες εκτός από τη δικαιοσύνη που είναι υπαριθμόν δύο η μεταρρύθμιση της δημόσιας δίκης, καταπολέμηση της διαφθοράς, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ανθρώπινα δικαιώματα συμπαραμένου και του δικαιώματο στην ιδιοκτησία. Έχει κάνει σημαντικέ προόδου και προσπάθειε η Ελβανία, όχι ότι τα έχει τελειώσει όλα, αλλά η πιο εντατική περίοδος διαπραγματεύσεων και μεταρρυθμίσεων είναι μετά την ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα κεφάλαια και με τις άλλες χώρες έχουμε περάσει και 6 και 7 και 8 και 9 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό, στη δικαιοσύνη κλπ. Και αυτό είναι τμήμα της δουλειάς μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις πρόσφατα εξέδωσε μια στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ ε, μετέβη τέλη Φεβρουαρίου στην Αλβανία Ε, δήλωσε ε, ότι σοβαρά ε, εννοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλει να ενταχθεί η Αλβανία, αλλά τους είπε ότι επίσης δεν μπορείτε να πείτε όπως είστε, πρέπει να αλλάξει η χώρα, να εντείνετε τις προσπάθειές σας και τα λοιπά, πάντα στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Σε αυτή τη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ανακοίνωσε ότι στο μέλλον θα επικεντρωθεί σε έξι εμβληματικές πρωτοβουλίες που είναι η ψηφιακή ατζέντα, το κράτος δικαίου, ασφάλεια και μετανάστευση, ε, ε, θέματα συνδέσεων, αγωγών, ε, μεταφορών και ενέργειας, κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και τέλος συμφιλίωση και σχέση καλής γειτονίας. Γιατί πρόκειται για μια ολόκληρη περιφέρεια όπου στη δεκαετία του 90 είδαμε πάρα πολύ φρικτά πράγματα και πολέμους. Χρειάζεται λοιπόν συμφιλίωση και σχέση καλής γειτονίας έτσι ώστε να αποφύγουμε χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκβιάζουν άλλες χώρες που θέλουν να ενταχθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να εισαγάγει στους κόλπους της διμερείς συγκρούσεις. Πρέπει αυτά τα θέματα να έχουν επιληθεί πριν ενταχθεί η χώρα. Η κυρία Μογκερίνη ήταν εκεί την περασμένη εβδομάδα για να ανακοινώσει αυτή τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τούτη τη εβδομάδα είναι και ο πρόεδρος Τούσκ. Πήγε και ο κύριος Γιούνκερ. Είναι η καιρή πάρα πολύ ε, φορτωμένη και στις 9 ε, Μαΐου που είναι η μέρα της Ευρώπης έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στην Αλβανία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας. Ε, το πρόγραμμά σας είναι πολύ καλό μείγμα, δείχνει όλες τις πτυχές του προγράμματος. Στα τύρανα θα δείτε ας πούμε και ένα εργαστήριο για την ασφάλεια των τροφίμων. Ε, θα δείτε την ε, Διεθνή Επιτροπή που ελέγχει τους δικαστές στον Αυλώνα στην Αυλώνα επίσης θα δείτε κάποιες ε, ε, εργασιακές συνθήκες. Έχουμε ε, θέματα που έχουν να κάνουν με δημόσιες προμήθειες, έμεση διαχείριση. Μόνο το 5% των διαγωνισμών και των προμηθειών διαχειρίζεται η ίδια η Αλβανία, αλλά θα δείτε και τα προγράμματα υποστήριξης του προπολογισμού τους. Ε, στην Αυλώνα θα δείτε και ε, ε, τη θάλασσα, τη παραλία, τα τουριστικά project. Υπάρχει και ένα έργο μεταφορών, είναι λίγο δύσκολο. Έχει ανανεωθεί ο διαγωνισμός, υπάρχουν προβλήματα, θα τα δείτε επιτόπου στην Αυλώνα όλα αυτά. Αυτά τα πέντε project λοιπόν που θα επισκεφτείτε νομίζω θα σας δώσουν μια εικόνα πλήρη και πραγματικά προσβλέπω στην επίσκεψή σας στην Αλβανία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κρίμα που δεν μπορώ να πάω. Είναι σημαντική η χώρα αυτή η Αλβανία πιστεύω και εγώ. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ποια ε, είναι η περιφερειακή συνεργασία ε, στα Βαλκάνια, πώς συνεργάζεται η Αλβανία με τις γειτονικές της χώρες εκεί στην περιοχή. Αναφερθήκατε σε αυτό για τις πρωτοβουλίες, το βρίσκω πάρα πολύ αξιέπαινο και αξιοσημείωτο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τελειοποιήσει ε, τις μεθόδους τους. Το τμήμα <laughs> διδάγματα από το, την εμπειρία έχετε κάνει μεγάλες ε, προσπάθειες και επιτυχίες. Υπάρχει μηχανισμός συνεργασίας και ε, ένταξης στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, που είναι οι δύο τελευταίες χώρες που μπήκαν. Υπάρχει αντίστοιχος ε, μηχανισμός για την Αλβανία, γιατί ήταν μέγα σφάλμα που δεν έγινε με την Κροατία. Ε, υπάρχει τέτοια συνεργασία οικονομική και γενικότερη, πώς το βλέπουν, γιατί οι χώρες που απεχθάνονται η μία την άλλη και δεν ανέχονται η μία την άλλη, εισάγουν ε, τις συγκρούσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουμε τώρα ανάγκη να εισάγουμε νέες συγκρούσεις. Αυτό έχει να κάνει και με τις οικονομικές σχέσεις και τα λοιπά. Ασχολούνται τα κράτη με αυτά. Υπάρχουν ε, ευρωπαϊκά κονδύλια που να ε, πηγαίνουν εκεί ή να μην πηγαίνουν. Μας απασχολεί αυτό το θέμα, μας τα αλανίζει. Δεν ξέρω αν έχουν ε, Άλλοι συνάδελφοι, ερωτήσει, όχι. Όλοι τα mail τους διαβάζουν. Ο κύριο Πυρίνσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δύο σύντομες ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Η μία ερώτηση αφορά ε, με τα περιφερειακά προγράμματα. Αναρωτιέμαι εάν ε, επιβλέπετε, παρακολουθείτε καθόλου τον διάδρομο ε, μεταφορών ε, που, έχει, που συζητιέται τα τελευταία 20 χρόνια είναι ο, διάδρομος ο νούμερο ε, περιθμών 8 μυθικών διαστάσεων η συζήτηση που θα φτάνει από, την, από τον Εύξηνο Πόντο μέχρι την Αδριατική. Ε, έχουμε δει ε, ότι υπάρχουν προβλήματα και με την ΦΥΡΟΜ, γιατί υπάρχουν προβλήματα εκεί με την ονομασία της χώρας. Αλλά ερωτώ, είναι κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο να συζητηθεί και να υπογραμμιστεί, μια και ανοίγει πλέον μια νέα διάσταση ε, για διασύνδεση Ανατολής Δύσης ή Δύσης Ανατολής αν προτιμάτε. Ανοίγονται κοινές δυνατότητες. Δεύτερη ερώτηση. Σχετικά με, την, ε, με τις CVM με το κράτος δικαίου και με την διαφθορά. Όταν μελετάτε τα θέματα αυτά στην περίπτωση της Αλβανίας, μέχρι ποιο βαθμό λαμβάνετε υπόψη τις διασυνοριακές ε, επιρροές. Γιατί ένα μεγάλο μέρος της διαφθοράς και οι εγκληματικές οργανώσεις δεν ε, περιορίζονται στην αλβανική επικράτεια, αλλά αποτελούν ε, πολύ καλά διακτηνισμένες εγκληματικές οργανώσεις από χώρες που αρχικά έχουν γεννήσει αυτή την παραβατικότητα. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, η περιφερειακή διάσταση και συνεργασία αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν. Ήδη στην ε, Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης άμα το σκεφτείτε, άμα το συγκρίνετε και με τη συμφωνία για την Ευρώπη, με την Ουγγαρία και την Πολυνία κτλ. λοιπά που είχαν συναυθεί, φαίνεται εδώ ότι αυτή η περιφερειακή συνεργασία πραγματικά της αποδίδεται μεγάλη σημασία από την αρχή. Τώρα ξανατονίζουμε αυτήν τη διάσταση ακόμη περισσότερο και αναφέρομαι και σας ε, ενημερώνω και για την ε, συνδιάσκεψη της ε, Σόφιας που θα γίνει το Μάιο υπό την αιγίδα της Βουλγαρικής Προεδρίας που είναι πρώτη φορά που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν με τους έξι αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των ε, Δυτικών Βαλκανίων. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που θα, που θα γίνει μια τέτοια συνάντηση. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και δραστηριοποίηση στα Δυτικά Βαλκάνια. Τους προσφέρουμε και τους παρέχουμε διαρκώς νέες ιδέες, κατευθύνσεις. Βεβαίως την ευθύνη ε, όλων αυτών θα την έχουν οι ίδιες οι χώρες. Δηλαδή να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές πριν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των ειδών. Ε, πρέπει λοιπόν από, πριν από την ένταξή τους να υπάρχει και μια αμοιβαία αναγνώριση δεξιοτήτων προσόντων προκειμένου να υπάρχει και ροή εργατικού δυναμικού από τη μία χώρα στην άλλη. Επίσης διοργανώνουμε και ανταλλαγές ε, αξιωματούχων κρατικών. Δηλαδή Αλβανοί ε, κρατικοί αξιωματούχοι πηγαίνουν στη Σερβία και το αντίστροφο κτλ. Και αυτό βοηθάει στην, ε, στη φιλίωση των κρατών αυτών. Και τέλος, κάτι ενδιαφέρον ενδεχομένως για την Αλβανία. Ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει αυτή η περιφερειακή ε, διάσταση, εκεί είναι η, η έδρα στα Τύρανα ε, και του Ευρωπαϊκού Γραφείου νεολαία. κατά τα πρότυπα ανταλλαγών νεολαία που, που διοργανώνονταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεταξύ Γαλλία, Γερμανία, Γερμανία, Πολωνία κτλ. κτλ. Και στα Δυτικά Βαλκάνια λοιπόν πλέον υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Και πρέπει να σας πω ότι και οι κρατικές αρχές, οι κυβερνητικές αρχές ε, ε, επιδεικνύουν μεγάλη δραστηριοποίηση στο Δυράχιο Πέρσι ε, διοργανώθηκε και μια σχετική συνδιάσκεψη και όλα αυτά βεβαίως ξέρετε έχουν αλλάξει και την ατμόσφαιρα, το κλίμα. Γιατί προφανώς ξέρετε ότι υπάρχουν εντάσεις μεταξύ Ελβανίας, Σερβίας, λόγω του Κωσυφοπεδίου για παράδειγμα αλλά παρόλα αυτά, για, αυτόν μάλλον το λόγο, είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν αυτές οι προσπάθειες. Για τον διάδρομο 8 το εξετάζουμε ακόμα. Βρισκόμαστε εμείς ε, έχουμε επικέντρωση των προσπαθειών μας στη μονάδα μου σε συγκεκριμένα θέματα. Πρέπει λοιπόν να ε, το δω και με τους συναδέλφους για να σας απαντήσω ολοκληρωμένα. Υπάρχει βεβαίως και μια μονάδα η οποία αφορά όλα τα, τα Δυτικά Βαλκάνια. Η δική μου μονάδα ασχολείται πιο πολύ με την Αλβανία. Βεβαίως όμως να το δω και να το συζητήσω και με τους συναδέλφους και να επανέλθω σε εσάς ε, έστω και διμερώς αν θέλετε για να σας ενημερώσω. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Να επιμείνω σε ένα σημείο θα ήθελα. Η φήμη της Αλβανίας είναι μία από τις χειρότερες, για να μην πω η χειρότερη, στον, ε, στους Ευρωπαίους. Το ξέρουμε από όλες τις έρευνες αυτό. Τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ένταξη της χώρας αυτής, ακόμα και για την προσέγγιση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν ξέρω, μισή, έξι μήνες πριν από τις ευρωεκλογές πραγματικά πρέπει να μας χαροποιήσει αυτή η συνδιάσκεψη στη Σόφια ε, και για τη συνδιάσκεψη με τα Δυτικά Βαλκάνια δεν ξέρω, χτυπάει λίγο η καρδιά μου με αυτά. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς μόνο να υπόσχεσαι ότι θα εντάξει τον άλλον. Πρέπει να κάνεις και απτά βήματα ε, και βεβαίως είναι προς το συμφέρον ολόκληρης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι χώρες να κάνουν βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως ταυτόχρονα σημειώνω και ε, την ε, ευρύτατη διαφωνία και δυσαρέσκεια των ευρωπαϊκών λαών όσον αφορά την προσχώρηση αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω ότι τα, προβλήματα είναι σύνθετα και χρειάζονται προσοχή, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε πραγματικά αξιόπιστε διαδικασίε. Δεν γίνεται να ξαναγίνουν εκπτώσει, ούτε να διευκολύνουμε ε, συγκεκριμένε χώρε, ακριβώ γιατί δεν μπορεί κανείς μόνο να υπόσχεται ή να διαπραγματεύεται. Υπάρχει λοιπόν κάποια, κάποιο σχεδιασμό για το πώς θα βελτιωθεί η φήμη της Αλβανίας στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί φαντάζομαι μια διαφημιστική εκστατεία δεν αρκεί. Απάντηση από την Κομισιόν. Ναι, ξέρετε ότι ξεκινάνε η διαδικασία σε ένταξη, ότι ανοίγει δηλαδή η διαδικασία ένταξη, δεν σημαίνει ότι αύριο εντάσσεται η χώρα. Ε, σημαίνει απλώς ότι θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τις απαιτήσει μας. Και πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι μακροχρόνια και αυτό είναι σαφές. Μόσο μόνο βέβαια μέσα από αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις ε, που θα πρέπει να τις κάνουν οι ίδιοι οι Αλβανοί, η ίδια η κυβέρνηση, έτσι ώστε να δείξουν ότι πραγματικά προσφέρουν αξιοπιστία, ε, μόνοι τους μπορούν να αντιστρέψουν αυτήν την κακή φήμη που ορθώς λέτε ότι υπάρχει όσον αφορά την Αλβανία. Μόνο μέσω των αποτελεσμάτων ε, μπορεί να αντιμετωπιστεί, να χτυπηθεί αυτή η εικόνα. Ε, αυτό που ε, ε, διαπιστώνουμε εμείς είναι ότι υπάρχει σαφής βούληση της κυβέρνησης της Αλβανίας να ε, ε, κάνει μεταρρυθμίσεις ε, και θα το δείτε και εσείς επί τόπου. Μας ζητούν οι ίδιοι να κάνουμε την επιτήρηση, το monitoring. Πραγματικά είναι η μοναδική χώρα που από μόνη της ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα, να, οι διεθνείς παρατηρητές να είναι παρόντες, έτσι ώστε να βλέπουν τους φακέλους των δικαστών. Επίσης, ε, ε, επέτρεψαν στην Guardia di Finanza ε, από την Ιταλία να φωτογραφίσει στην ουσία ολόκληρη τη χώρα ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να φωτογραφίσουν. Καμία άλλη χώρα δεν θα επέτρεπε ε, ε, ελεύθερη πρόσβαση στον εναέριο χώρο της ε, και ελευθερία να πάρει μια άλλη χώρα όποιες φωτογραφίες θέλει. Αυτό σημαίνει ότι μας δίνουν την δυνατότητα, μας επιτρέπουν να δούμε, να παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά το τι κάνουν και φαίνεται ότι υπάρχει από τη μεριά τους η βούληση να κάνουν κάτι. Επίσης φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό έχουν υπάρξει πολλές κατασχέσεις ε, ναρκωτικών και λοιπά. Φυσικά δεν εξαντλείται έτσι με αυτό η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν και παρακλάδια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να το χτυπήσουμε. Αλλά και αυτό είναι ένα τμήμα της ε, συνεργασίας. Έχουμε επίσης ε, και ε, ε, αξιωματικούς σύνδεσης liaison officers της Europol άρα συνεργασία και με την Europol. Ε, επομένως λέω ότι ε, εντα, εντείνεται ε, προς την σωστή τροχιά και κατεύθυνση η συνεργασία. Το γεγονός πάντως παραμένει ότι πρέπει να πείσουμε την κοινή γνώμη, τον κόσμο, μέσω των αποτελεσμάτων, μέσω συγκεκριμένων αξιόπιστων αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν θυμάμαι καλά, γιατί ε, ασχολούμαι με ε, διευρυνσει ε, εδώ και 20 χρόνια και μπορώ να σας πω ότι όταν η Πολωνία ξεκίνησε τον μακρύ της δρόμο που την οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ε, προκαταλήψεις ήταν πάρα πολλές, πολλά και τα ε, δίθεν αστιάκια, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, τα ακούσατε κι εσείς στη γερμανική τηλεόραση. Εδώ δεν αναφέρομαι σε πολιτική κατάσταση, αναφέρομαι σε όλα τα υπόλοιπα, στην ιδέα που έχουν οι άλλοι για τη χώρα κτλ. Ε, και βεβαίως η χώρα πλέον, η Πολωνία, έχει μια εντελώς διαφορετική φήμη σήμερα. Πολύς και μακρύς ο δρόμος, ε, είναι γεγονός πάντως ότι η αλβανική πλευρά θέλει να μπει στην επόμενη διαδικασία έτσι ώστε και υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποχρεωθεί ε, να ε, κάνει τα πράγματα σωστά όσον αφορά την Αλβανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι οπωσδήποτε η ώρα να πάμε εκεί. Η πρώτη φορά από τότε που έχω αίσθηση εδώ για την Επιτροπή, οι συνάδελφοι Βον Μαρινέσκου, Τσανέσκι και κλίν θα πάνε. Ο κύριος Βάλλη ε, απέσυρε τη συμμετοχή του σήμερα το πρωί. Ζητούνται και άλλοι εθελοντές γιατί τη σημαντική αυτή αποστολή. προσπάθησε χτες να ε, πείσω τον συνάδελφο Άσουαρθ, αλλά δεν ψήνεται. Όλοι έχουν δικαιολογίες γιατί δεν μπορούν να πάνε. Θα παραμείνουμε σε επαφή οπωσδήποτε και σας ευχαριστώ. Και φτάσαμε στο σημείο 5, ε, η ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του 2018 για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων κινητικότητα των εργαζομένων σημαντικό θέμα γιατί έχουμε σήμερα ψηφοφορίες σε άλλες ε, επιτροπές για την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Ο κύριος Πυρίνσκι εκπροσωπεί την εισηγήτρια και ο κύριος Πούφαν, τον οποίο καλωσορίζω θερμά, έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Για τα καλά σας λόγια και για το λόγο που μου δίνετε. Καλημέρα σε όλους σας, κυρίες και κύριοι. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε την πέμπτη πεντηκοστή επέτειο ε, για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Σε όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι εργαζόμενοι χωρίς διακρίσεις με βάση την εθνικότητα ε, για τους όρους εργασίας, την αμοιβή τους κλπ. Το 2015 11,3 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών εργάζονται και διαμένουν σε διαφορετική χώρα μέλος από την πατρίδα τους. Ε, αυτά τα στοιχεία ε, αντιστοιχούν στο 3,7% του συνόλου του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε ε, ηλικία που μπορεί να εργάζεται. Σε ό,τι αφορά τις ροές των πολιτών αυτό, 1,1 εκατομμύριο το 2014 άλλαξαν κράτος μέλος. Άλλο 1,3 εκατομμύριο ε, διασχίζουν ε, ε, συνήθως σύνορα για να εργαστούν σε διαφορετική χώρα από εκείνη που διαμένουν. Ε, οι δικές μας εργασίες ε, σε τι συνίστανται για την έκθεση αυτή. Για την έκθεση για την κινητικότητα των εργαζομένων αξιολογήσαμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγυάται την ελευθερία της κυκλοφορίας και έχουμε αξιολογήσει τις δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση της κινητικότητας. Από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 2017 αναλύσαμε τα ενημερωτικά μέσα και εργαλεία που παρέχει στους εργαζομένους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκείνους που ε, εξετάζουν το εδεχόμενο να εγκατασταθούν σε ε, άλλο κράτος μέλος και ε, πώς δαπανώνται τα κονδύλια από το πρόγραμμα EASY και το Κοινωνικό Ταμείο. Για την ενίσχυση στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 et avons examiné ε, υπάρχουν διασυνοριακοί ε, εργαζόμενοι που καλύπτονται από το Γιούρες και ε, άλλα προγράμματα το 2016 και 2015. Εκτός από το λογιστικό έλεγχο, κάναμε έλεγχο για τη λειτουργία του δικτύου EURES και τέλος αναλύσαμε και την ποιότητα ενός δείγματος ε, ε, θέσης ε, εργασίας, αγγελίας στο EURES, στη σελίδα αυτή, στη δικτυακή πύλη έχει δημιουργήσει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Solvit, το Eures και το, η Ευρώπη είναι δική σας για να διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων και τα κράτη-μέλη τα ίδια έχουν ενημερωτικά site για να ενημερώνουν τους εργαζόμενους από τις άλλες χώρες που εργάζονται στην επικράτειά τους ή τους ίδιους πολίτες τους που θέλουν να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν διαθέτει πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλουν κάθε διάκριση αντίθετη με την ελευθερία της κυκλοφορίας. Εκτός από αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει τις ε, περιπτώσεις και τις υποθέσεις που έχουν ε, ε, για τις οποίες έχουν προσφύγει στα κράτη-μέλη, γιατί δεν ενημερώνεται συστηματικά, δεν κοινοποιούνται. Υπάρχουν ε, και κάποια εμπόδια που μπορεί να μην ε, συνιστούν παραβίαση δικαιωμάτων των εργαζομένων, παρόλα αυτά ε, δέχεται να εμποδίσουν την κινητικότητά τους, όπως είναι η μη αναγνώριση των προσόντων και των δεξιοτήτων, το πρόβλημα της γλώσσας ή η μη δυνατότητα μεταφοράς θεμελιωμένων δικαιωμάτων ε, συνταξιοδοτικών κλπ. Το 2014 έγιναν διάφορες μελέτες που έδειξαν ότι γύρω στα 2,9 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών θα επιθυμούσαν να έχουν μεταβεί και να κατασταθούν το 2015 σε άλλο κράτος μέλος. Αλλά πάνω από ένα εκατομμύριο περίπου κατάφεραν να το κάνουν αυτό. Άρα υπάρχει πρόβλημα ε, για τη γνώση των δράσεων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διευκόλυνση της κινητικότητας στη σημερινή προγραμματική περίοδο 2014-2020 τα κράτη-μέλη είχαν τη δυνατότητα να αντλήσουν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα προγράμματα και τις περιόδους άσκησης και μαθητείας στάζ σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Το 2013 και 2014 όταν εγκρίθηκαν τα διάφορα ε, ΕΣΠΑ και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήλεγξε ε, αν ήταν σε θέση τα κράτη-μέλη, αν είχαν προγραμματίσει τέτοιες δράσεις υπέρ της κινητικότητας των εργαζομένων. Και δεν ξέρουμε ε, εάν άντλησαν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η βασική πηγή χρηματοδότησης λοιπόν ε, παραμένει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την, την, την, την ε, ε, κοινωνική καινοτομία, το EASY, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 23 διασυνοριακά προγράμματα έχουμε μελετήσει, Γιούρες και EASY. Λίγα είναι τα έργα που έχουν καλά αποτελέσματα. Ας πούμε, ο αριθμός των ανέργων που αναζητούσαν εργασία και βρήκαν δουλειά. Το πρόγραμμα εμφανίζει προβλήματα και ανεπάρκειες. Το βασικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι αυτό για τη διευκόλυνση των ε, εργαζομένων, αλλά δεν δημοσιεύονται αυτά πάντα σε εθνικό επίπεδο, οι προσφορές δηλαδή. Ε, μπορεί οι προσφορές να είναι στη διαδικτυακή πύλη, αλλά δεν περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για εκείνους που ζητούν εργασία, όπως είναι ε, ο μισθός ή η προθεσμία κατάθεση υποψηφιοτήτων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν γίνει αποσπάσεις περίπου 30.000 ε, το 2015 από το Γιούρες που σημαίνει μόνο 3,7% των ε, επαφών μεταξύ ε, των συμβούλων του Γιούρες και των υποψηφίων εργαζομένων. Δεν είναι πολύ γνωστά τα εργαλεία που διευκολύνουν την κυκλοφορία των εργαζομένων ή ε, που τους επιτρέπουν να καταγγείλουν διακρίσεις. Αντίστοιχα και τα στοιχεία για τις ροές των εργαζομένων, για το είδος της δουλειάς, για τις ε, ανισορροπίες στην αγορά εργασίας. Πρέπει να βελτιωθούν οι μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κινητικότητα των εργαζομένων για να υπάρχει εξασφαλισμένη συμπροματικότητα και καλύτερη παρακολούθηση των επιδόσεών τους. Το Γιούρις και το Ίζι πρέπει να βελτιωθούν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων για να, υπάρχει, ε, να γίνει ένα γνήσιο εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόσληψη και την τοποθέτηση των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς. Ο συνάδελφος Πυρίνσκι έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως σημειώσατε κι εσείς, είναι ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και απασχολεί τις συζητήσεις μας συχνά. Η συγγήτρια θα ήθελε να σημειώσει τα εξής. Η έκθεση που παρουσίασε το συνέδριο είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Πουφάν και το επιτελείο του αξίζουν συγχαρητήρια για το έργο τους και ιδίως για το γεγονός ότι οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις τους δεν αφορούν μόνο την ε, αξιοποίηση δημόσιων κονδυλίων, αλλά αποδίδουν τη δέουσα σημασία στον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν αυτή τη θεμελιώδη ελευθερία. Γίνεται προφανές από τα πορίσματα του συνεδρίου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και προκλήσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία που πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τους Ευρωπαίους συνομοθέτες, όπως για παράδειγμα η κατάργηση εμποδίων για την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, και ε, προκειμένου να καταστεί η διαδικασία αυτή απλή, φιλική προς το χρήστη, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις δημόσιες διοικήσεις η άλλη, μια άλλη παρατήρηση του συνεδρίου είναι η ανάγκη καλύτερου συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ιδίω όσον αφορά τη συμπληρωματική ασφάλιση και τα καθεστώτα, προκειμένου να ε, καταργηθούν αντικίνητρα για την κυκλοφορία των εργαζομένων. Είναι υποχρέωση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει υπόψη της τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υποβάλει σχετικές προτάσεις, απαντώντας σε αυτές. Μεταξύ άλλων θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση αναφέρεται και ένα πρόβλημα σχετικά με την ε, ε, ε υλοποίηση διασυνοριακών προγραμμάτων για την απασχόληση. Η Κομισιόν και ιδίω η Γενική Διεύθυνση Απασχόληση πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα στην επόμενη πρόσκληση υποβολή προτάσεων και να εντάξει υποχρεωτικά κριτήρια αποτελεσμάτων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων προκειμένου να μετράτε στην πράξη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και τα σχόλια που παραλαμβάνει. Επίσης, η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης πρέπει να συντάξει κατευθύντριες γραμμές για τους συντονιστές γιούρες, τους εθνικούς συντονιστές, και τις αρχές έβρεσης εργασίας και ε, την ε, ανάγκη ε, συνδυασμού όλων των ταμείων. Πρέπει επίσης οι διαχειριστικές επιτροπές των κρατών μελών να αξιοποιούν ε, σε μεγαλύτερο βαθμό ε, τις δυνατότητες που δίνει το ESF και τα προγράμματά του. Αυτές οι ευκαιρίες και δυνατότητες μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν αναντιστοιχίες μεταξύ προσόντων και ελλείψεις ε, εργατικού δυναμικού. Η ελεύθερη, η ελεύθερη κυκλοφορία λοιπόν είναι ε, βασικό στοιχείο της ενιαία αγοράς, όμω φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για τη δημιουργία μιας πραγματικής γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασία. Η αξιοποίηση λοιπόν του EURES ε, ως ένα εργαλείο που θα είναι προσβάσιμο σε όλα τα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντική Φαίνεται όμως ότι κάποια κράτη-μέλη ε, ε, ε, δημοσιεύουν στην πύλη αυτή μόνο κάποιες από, από τις θέσεις εργασίας. Κάποιες χώρες, όπως οι κάτω χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία, κυμαίνονται σε ποσοστά δημοσίευσης κενών θέσεων από το 9% στο 16%, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες πραγματικά δημοσιεύονται όλες ενώ σε κάποιες χώρες ε, άλλες ε, μειώθηκε και το ποσοστό κάτω από το 50% το 2016 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Επίσης, το συνέδριο εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την ποιότητα των κενών θέσεων που δημοσιεύονται στο πόρταλ, καθώς 39 από τις 50 θέσεις ε, που εξετάστηκαν δεν περιείχαν σημαντικέ πληροφορίε όπω για παράδειγμα η προσωρινή καταβολή υποψηφιωτήτων. Αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την ε, Κομισιόν και από τι αρχέ των κρατών μελών ε, ευθυγραμμισμένα με την σύσταση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου προκειμένου το γύρω να γίνει ένα πραγματικό ευρωπαϊκό εργαλείο. Εντόπισε λοιπόν το συνέδριο μέσα από προβλήματα τα οποία πρέπει και ζητούν άμεση δράση από τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν προκειμένου να προωθηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων και να δημιουργηθεί μια γνήσια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Κατ' εξαίρεση θα δώσω το λόγο και σε ένα μέλος του Μαρτίνα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ το ελεγκτικό συνέδριο για την εργασία τους. Όπως είπατε Κύριε Πρόεδρε, θα γίνει και μια ψηφοφορία σήμερα στην Επιτροπή Απασχόλησης που θα αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας και το νομίζω ότι συνδέεται πάρα πολύ με όλα τα θέματα τα οποία συζητούμε τώρα, με τη δέσμη κινητικότητας, τους μετα ε, τους αποσπασμένους εργαζόμενους κτλ. Ε, η ελευθερία κυκλοφορίας λοιπόν ε, για τους πολίτες αποτελεί ακρογωνία ολίθο της ενωσιακής ηθαγένειας και σαφώς αναφέρεται ρητά στις συνθήκες. Περίπου 4% του εργασιακού δυναμικού σε ηλικία απασχόλησης μετακινείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι ε, πιο ε, υψηλό γιατί το ποσοστό κινητικότητάς μας σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 10 φορές μικρότερο βεβαίως διαφέρουν και οι καταστάσεις. Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν προσκόμματα ε, κυρίως για τους μακροχρόνιους ανέργους και νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να γνωρίσουν οι πολίτες τα σημερινά και μελλοντικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να βοηθηθούν. Ε, η κινητικότητα μπορεί να μειώσει πολύ την ανεργία, κυρίως δε την ανεργία των νέων γιατί σε ορισμένες ε, περιοχές έχουμε νεανική ανεργία του 50% ενώ υπάρχουν ε, άλλες περιφέρειες όπως ας πούμε στη δικιά μου χώρα όπου το ποσοστό απασχόλησης των νέων είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτόν τον μεγάλο σκόπελο της αναντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά τις ειδικότητε Νομίζω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε περισσότερο αυτά. Είδα τα αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων ε, ε, σύμφωνα με την χώρα και με προβληματίζει το γεγονός ότι η περισσότερη το περισσότερο ποσοστό κινητικότητας ε, προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και ακριβώς αυτοί είναι που θα υποφέρουν περισσότερο, είναι πιο ευάλωτοι απέναντι στο Brexit. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Κάτι άλλο. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπατε, δεν έχει αρκετές πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κινητικότητα των εργαζομένων και δεν πράττει ε, τα κατάλληλα έτσι ώστε ε, να προχωρήσει στην αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων και δεξιοτήτων. Πού είναι το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα δεδομένων, είναι πρόβλημα στάσης, είναι πρόβλημα ανταλλαγής πληροφοριών, προέρχεται το πρόβλημα από τα κράτη-μέλη κυρίως. Επίσης, όσον αφορά ε, τι, τι, προβλέπει η Κομισιόν όσον αφορά τα, το επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα δημοσιευθεί τον Μάιο, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Και τέλο, αλλά εξίσου σημαντικό, από άποψη ελέγχου του προπολογισμού, ξέρετε ότι η αποτελεσματικότητα της χρήση των πόρων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Μιλάμε διαρκώ και όλο και περισσότερο για ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ε, των ε, δαπανηθέντων ε, ευρωπαϊκών πόρων πώς μπορούμε να δείξουμε ε, στην πράξη ε, μέσω της κινητικότητας στους ε, Ευρωπαίους πολίτες αυτή την αποτελεσματικότητα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη ερώτηση έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο για την έκθεση καταρχάς. Σε σχέση με αυτό, ε, είχα κάποια ε, συνομιλία ε, με τον υπεύθυνο της διασυνοριακής περιοχής Γιου Ρέγγιο Μας Ρήνου, το δύο ποταμών με Ρήνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός, αλλά είναι ένας άνθρωπος. Πώς θα υποστηριχθούν αυτές οι θέσεις ενημέρωσης και παροχής συμβουλών του Γιούρες οι οποίες ε, υποχωρούν. Πώς μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τις ενισχύσει και να υπάρχει και καλύτερη πρικοδότηση, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή οι διαμεσολαβητές. Ο συνάδελφος Άσχουρτ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να υποστηρίξω αυτό που υπόθηκε νωρίτερα σχετικά με την έλλειψη δημόσιων πληροφοριών και στοιχείων. Εγώ, ναι, είμαι Βρετανός όπου η κοινωτικότητα των εργαζομένων έχει επιφέρει σημαντικότατα ωφέλη στην οικονομία. Και αυτό είναι προφανές παντού, αλλά πρόκειται για μια χώρα όπου η κυκλοφορία εργαζομένων ήταν πολύ ακαθόντες θέμα. Η μεγαλύτερη συζήτηση και διαμάχη, διαφωνία βασίστηκε σε πεπιθήσεις που διαψεύστηκαν από την πραγματικότητα υπήρξε για παράδειγμα μια δημόσια συζήτηση ότι η κυκλοφορία εργαζομένων θα επιτρέψει σε εργαζόμενους από το εξωτερικό να έρθουν και να μειώσουν τους μισθούς. Εγώ ε, είχα πει στους ε, ε υπαλλήλου του ελεκτικού συνεδρίου ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό. Είναι γεγονός ότι οι ε, εργαζόμενοι ε, χαμηλών προσόντων ε, μπορεί να, ε, να είναι πιο ορατή ε, και να τους αφορά αυτό σε ένα μεγαλύτερο βαθμό, αλλά δεν αφορά τραπεζίτες γιατρούς. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, πρόσβαση στις, στις, στα κοινωνικά επιδόματα. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα που συνδέεται πολύ συχνά με, με τη συζήτηση αυτή. Άρα, θεωρεί το ελεγκτικό συνέδριο ότι η Κομισιόν απέτυχε να δημοσιεύσει αυτά τα στοιχεία, αυτές τις πληροφορίες και κατά τον τρόπο αυτόν ε, έθεσε μήπως σε κίνδυνο την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ ο κύριος Ζαντών για την Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια, για τις ερωτήσεις. Ξέρετε ότι Συνήθως ευχαριστούμε το ελληνικό συνέδριο λοιπά. Λόγω του έργου όμως και των συζητήσεων που είχαμε την ε, τελευταία χρονιά, πράγματι είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες ε, συζητήσεις και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Και γι' αυτό και αποδεχόμαστε όλες τις συστάσεις και το βλέπετε και στην πράξη αυτό. Θέλω να επιμείνω σε τρία θέματα. Πρώτον, για το ίδιο το θέμα της συστάσεις και τρίτον, για τα βασικά διδάγματα που αντλούμε από την ε, διαδικασία αυτή. Υπόθηκαν και από άλλους, οπότε δεν θα τα επαναλάβω, αλλά είναι προφανές ότι μιλάμε για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων ως ε, θεμελιώδη αξία και πυλώνα ε, του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Και συγκεκριμένα μιλούμε για τη δυνατότητα των Ευρωπαίων πολιτών, των εργαζομένων, να ε, εγκαθίστανται και να εργάζονται και να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή οποιοδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από ορισμένες εβδομάδες, ενδεχομένως ε, είδατε, διαβάσατε μια έκθεση, ετήσια έκθεση, για την κινητικότητα των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην έκθεση αυτή υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, πληροφορίες, σχετικά με τους ε, ε, μετακινούμενους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιοι είναι, από πού κατάγονται, από ποιες χώρες προέρχονται, προς τα πού πηγαίνουν. Δείτε την αυτή την έκθεση γιατί πραγματικά είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Και ακριβώς επειδή αφορούσε και το 2017, ε, είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία επιβεβαιώνει και κάποιες τάσεις που είχαμε διαπιστώσει ε, και νωρίτερα ε, σύμφωνα με τις οποίες, ότι, ε, σύμφωνα με, την, με η κινητικότητα των εργαζομένων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται. Το συνέδριο αναφέρεται σε 11 εκατομμύρια, εμείς μιλούμε για 17 εκατομμύρια αν συνυπολογίσεις και τους συνταξιούχους και τις οικογένειες των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 17 εκατομμύρια πολίτες που έχουν κάνει αυτή την επιλογή, ξέρετε, να μετακινηθούν, να μετακομίσουν σε, σε ένα άλλο κράτος μέλος. Ε, βλέπουμε την ίδια τάση και για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Αν συγκρίνουμε τα στοιχεία με, με δεκαετίες, με τα στοιχεία, ε, η τάση ε, είναι αντίστοιχη από 1,3 εκατομμύρια σε 2,4 αν τα θυμάμαι σωστά. Το ίδιο και για τους εργαζόμενους που μετακινούνται από τη μία πόλη στην άλλη χρησιμοποιώντας και διεθνείς μεταφορές. Υπάρχει παρόμοια τάση. Πώς γίνεται αυτό Μα ακολουθούμε πολιτική ε, διακρίσεων στη βάση της εθνικότητας, ε, έχουμε καταργήσει εμπόδια, έχουμε θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο, πολύ σημαντικό, έχουμε κανονισμούς, οδηγίες και θα έχετε δει ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια ε, υπήρξαν έντονες συζητήσεις για το νομικό αυτό πλαίσιο και με εσά εδώ, με, την ε, υιοθέτηση, με την έγκριση εκτελεξιστικών πράξεων, ε, και κανονισμών και ε, ελπίζω και με την βοήθειά σας ε, το Κοινοβούλιο θα συνενέσει και στην αναθεώρηση που ξεκίνησε το 2016. Έχουμε λοιπόν θεσμικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο, έχουμε και εργαλεία. Έχουμε εταιρικέ σχέσεις, έχουμε αξιωματικούς συνδέσμους, έχουμε το πόρταλ του Γιούρες έχουμε και προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν κάποια από τα έργα, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και φυσικά όλα αυτά διασυνδέονται. Τα, τα, τα εργαλεία που έχουμε και τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε πρέπει να αντικατοπτρίζουν βεβαίως τη φιλοδοξία που έχουμε. Ε, η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου αφορά ακριβώς αυτό το τελευταίο κομμάτι. Για τις συστάσεις. Εγώ θέλω να ξαναδούμε λίγο τον τίτλο της έκθεσης που θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει πλήρως τα βασικά μηνύματα του ελεκτικού συνέδριου. συνεδρίου. Ε, ελευθερία κυκλοφορία εργαζομένων, ε, θεμελιώδης αξία, αλλά χρειάζεται καλύτερη αξιοποίηση. Είναι λοιπόν μια σύσταση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τα κράτη-μέλη που βεβαίως διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτό. Ε, σε σχέση με ε, τις μετρήσεις που κάνουμε, πράγματι πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και να μετρήσουμε αν οι, ίδιοι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θεωρούν ότι έχουν ε, επαρκείς πόρους στη διάθεσή τους, αν η βοήθεια που λαμβάνουν είναι επαρκής. Ε, το Solvit, το Eures, όλα αυτά που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του, του, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Στο Solvit δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε γιατί αφορά άλλη, άλλη μονάδα της Κομισιόν. Αλλά για το ε, για την πύλη Γιούρες πραγματικά τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Είναι γεγονός. Ε, κάθε μήνα έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές στην πύλη Γιούρες και πάνω από 1,2 εκατομμύρια επισκέψεις. Βεβαίω, ε, υπάρχουν και περιθώρια βελτίωση και μπορεί και να πλουστευτεί η διαδικασία. Για τη σύσταση 2, την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών προκειμένου να εντοπίζονται ε, διακρίσει κατά τη ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό συνδέεται και με τη σύσταση 3 για την βελτίωση της συλλογής και αξιοποίησης ε, δεδομένων για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και την κινητικότητα των εργαζομένων. Συμφωνούμε απολύτως. Πρέπει να δούμε πώς θα βελτιωθούμε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν ε, ενέκρινε ε, την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής για την Απασχόληση και μάλιστα συνέστησε και μια ομάδα ε, εξειδικευμένη, η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση ε, κινδύνου και έχουμε κάνει και κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σύσταση 4. Βελτίωση της ε, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, του σχεδιασμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προτείνεται να ενισχυθούν οι συνέργειες και συμπράξεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του προγράμματος EASY. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, σε ένα βαθμό μπορούμε να το κάνουμε. Ε, το, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βρίσκεται υπό κοινή διαχείριση, το EASY υπό αποκλειστική διαχείριση. Εν πάση περιπτώσει, στις 2 Μαΐου θα υποβληθούν και σχετικές προτάσεις, όπως γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή εγώ δυσκολεύομαι, όπως καταλαβαίνετε καταλαβαίνετε να, να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή και του ζητά να ολοκληρώσει. Συστάσεις 5 και 6 για το πόρταλ ε, του Γιούρες και εδώ χάρη στην νομοθετική αρχή έχουμε κανονισμό που ενεκρίθη το 2016 με Έτοιμα να υπάρχει και ένας μηχανισμός αξιολόγησης επιδόσεων από τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή. Αυτό ενεκρίθη έπειτα από πολύ μακρές συζητήσεις με, το, τα κράτη-μέλη και πλέον βρισκόμαστε στη φάση εφαρμογής. Σκοπός μας είναι λοιπόν το, το EURES να καταστεί ένα πραγματικό ευρωπαϊκό εργαλείο και τέλος πρόταση για την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Απασχόλησης. Ξέρετε ότι αυτό σχετίζεται με τη βελτίωση τη ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώ και τη δυνατότητα των αρχών αυτών να ε, διαμεσολαβούν στον τομέα τη ε, κινητικότητα των εργαζομένων. Αυτά ε, ξέρετε ότι η έκθεση αυτή χρησιμοποιήθηκε και στην αιτιολογική έκθεση τη πρόταση αυτή και νομίζω ότι με όλα αυτά τα στοιχεία θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Σύντομη παρουσίαση σημαίνει ένα τέταρτο, 15 λεπτά Ενα πέντε. όχι 35. Συγγνώμη. Sorry. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σταματήσουμε και θα τον γράψουμε ξανά στην ημερήσια διάταξη σε μελλοντική φάση για ε, μεγαλύτερο βάθο συζήτηση. Damit sind wir am Ende Τελείωσε και το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Χρειάζεται λίγο άσκηση για να δούμε ποια είναι η σύντομη παρουσίαση και ποια όχι για να μάθουμε όλοι από όλα αυτά. Καλωσορίζω θερμά τον Υπουργό Οικονομικών της Ουκρανίας ε, και τη Γενική Διευθυνσία. Χαιρόμαστε που είστε εδώ κύριε Ντανίλιουκ. Ε, επανειλημμένα έχουμε ασχοληθεί με την Ουκρανία. Το Μάιο του 2016 είχαμε μεταβεί επίση στη χώρα και είχαμε και την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του 2016 για την Ουκρανία, ε, την οποία λάβαμε υπόψη. Και ε, χαρήκαμε που καταφέρετε να έρθετε. Θέλουμε μια ενημέρωση για την κατάσταση στην Ουκρανία και για την οικονομική βοήθεια φυσικά. 8 δισεκατομμύρια είναι οι επιδοτήσεις και 5 δις μακροοικονομική βοήθεια για τον προϋπολογισμό με τη μορφή δανείων μέχρι το έτος 2014-2015 μάλλον και έκτοτε από το 2014 και μετά Έχουμε μια νέα ε, συμφωνία, 11,2 δισεκατομμύρια και με πολλά δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Thank you. Good morning. Καλή σας μέρα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη μου τιμή που ε, είμαι σήμερα εδώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού έτσι ώστε να υποστηρίξω την πρωτοβουλία για την μακροοικονομική ε, ε, οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, MFA εφ' Παρά την τεράστια προσπάθεια ε, και πρόοδο όσον αφορά τις ε, πρόοδους ε, που κατεβλήθησαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εξεκολουθεί η Ουκρανία να βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και ε, λόγω της έλλειψης μεταρρυθμίσεων των ετών πριν από τον πόλεμο και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο χρόνο έτσι ώστε να μεταρρυθμίσουμε τη χώρα. Ας δούμε κάποια στοιχεία όσον αφορά το 2014, το 2015 ε, και την, σημερινή, κατάσταση έτσι όπως έχει σήμερα χάσαμε με τον πόλεμο 16% του ΑΕΠ. Ε, ο πληθωρισμός έφτασε στο 44% το έλλειμμα στο 5% ε, και ε, το απόθεμα των κεντρικών τραπεζών έφτασαν σε κρίσιμο χαμηλό επίπεδο, κρίσιμα χαμηλό επίπεδο. Επίσης, ε, ε, εξαρτώμαστε πλήρως από την Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά το φυσικό αέριο και το εμπόριο. Τέσσερα χρόνια μετά, επιστρέφουμε πλέον σε οικονομική ανάπτυξη με τίσιο ποσοστό 3%. Ο πληθωρισμός για φέτος θα είναι μονοψήφιος, περίπου 9%. Ε, μειώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα ε, σε 1,5% την προηγούμενη χρονιά και συνεχίζουμε ε, να ε, καταβάλουμε προσπάθειες σχετικά με το θέμα αυτό. Έχουμε αποκαταστήσει τις, τα αποθέματά μας που φτάνουν πλέον σε 19 δις δολάρια. Και προσπαθούμε βέβαια να διαφοροποιήσουμε και το εμπόριό μας. Και όλα αυτά τα επιτύχαμε λόγω των πολύ φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων που έχουμε προγραμματίσει, αλλά βεβαίως και από την βοήθεια που δεχόμαστε από την διεθνή κοινότητα, αλλά φυσικά ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια πετύχαμε περισσότερα από όσα είχαν επιτευχθεί στα 23 χρόνια της ανεξαρτησίας. Από τη στιγμή της ανεξαρτησίας δηλαδή μέχρι το ξεκίνημα του πολέμου. Ε, πολλές, ε, πολλές μεταρρυθμίσεις για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, για να βελτιώσουμε το σύστημα ε, μειοδοτικών διαγωνισμών για τη δικαιοσύνη, για την μεταρρύθμιση της υγείας. Κάναμε καθαρίσεις πολλές και εξηγιάναμε τον τραπεζικό τομέα κλπ. Αλλά βεβαίως δεν είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος των μεταρρυθμίσεων. Πολύ ε, μεταξύ ημών, ε, σκεπτόμενοι τα όσα έχουν συμβεί κατά διαστήματα στις χώρες σας, ε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις παίρνουν χρόνο. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ουκρανία. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε επιπρόσθετη βοήθεια έτσι ώστε να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και έτσι ώστε η οικονομική μας κατάσταση να ενισχυθεί για το τρέχον και επόμενο έτος, 18 και 19 ή έχουμε ένα ε, πρόβλημα όσον αφορά την ε, ε, εξισορρόπηση των κονδυλίων και όσον κυρίως προχωρώντας προς το 2020 έχουμε ένα εξωτερικό χρέος 7 δις, 4 όμως δις θα μπορούσαν να αναπληρωθούν από το εμπόριο και από το πρόγραμμα IMF τα υπόλοιπα από άλλες ε, συμβατικές ε, πηγές. Ε, και αυτό βεβαίως εξηγεί γιατί το μακροοικονομικό σύστημα είναι τόσο σημαντικό για μας. γιατί και, πόσο μπορεί να μας βοηθήσει μια τέτοια υποστήριξη, μια τέτοια βοήθεια. Πρέπει να γίνουν κατανοητές ε, οι τα διακυβεύματα, οι προκλήσεις που έχουμε, ε, γιατί εδώ βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, σε ένα σημείο καμπή. Ε, έχουμε και κάποια θεσμικά προβλήματα, τα οποία έχουν κληροδοτηθεί από το παρελθόν. Ε, έχουν συμβεί και σε άλλες χώρες και η Ουκρανία δεν είναι κάτι καινούριο. Εμείς ε, ε, αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία σε όλα αυτά τα θέματα και άλλωστε οι πρόοδοι των τεσσάρων τελευταίων ετών ε, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στίχημα αυτό. Έχουμε το, σύστημα, έχουμε το πρόβλημα ε, της, το δημογραφικό πρόβλημα. Έχουμε μεγάλη μείωση δημογραφική που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις εξελίξεις στη χώρα Έχουμε επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα κόπωσης ε, του πληθυσμού, ε, καθώς επίσης ε, και η κατάσταση με την Ρωσία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από καθαρά οικονομική άποψη όμως πρέπει να γνωρίζετε το εξής. 5% ή πάνω από 5% του ΑΕΠ μας κατευθύνεται στην άμυνα και την ασφάλεια είναι ε, το υψηλότερο ποσοστό απανταχού της γης. Παρόλες ε, τις ε, τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις, οι προκλήσεις είναι σημαντικές και οδηγούν την, το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων και περνούν βεβαίως από την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. κύριες πρωτοβουλίες ε, πλέον είναι να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις ε, που έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε περάσει πολλά νομοσχέδια, έχουμε δημιουργήσει ένα σημαντικό ε, πλαίσιο έτσι ώστε να μεταρρυθμιστούν και οι πιο σημαντικές περιοχές, οι πιο τα πιο σημαντικά πεδία και τώρα πρέπει βεβαίως να περάσουμε στην υλοποίηση και αυτό θα πάρει αρκετά χρόνια. Ε, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία αυτά ε, οι ιδιωτικοποιήσεις, ε, ο τομέας της ενέργειας, η καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω συγκεκριμένων υποδομών που δημιουργήθηκαν από μηδενική βάση στη χώρα μας. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και η τελειοποίηση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία ε, των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά τα οποία πλουτίζουν το θεματολογιό μας των μεταρρυθμίσεων. Ε, όσον αφορά το MFA. δεν έχουμε ολοκληρώσει όλες τις, ε, ε, τις, ε, όλα τα προαπαιτούμενα όσον αφορά το μακροοικονομικό σύστημα. Έχουμε λάβει 600 εκατομμύρια ευρώ. Um. Δεν λάβαμε άλλωστε τα 600 εκατομμύρια της τελευταίας δόσης και όσον αφορά τις προϋποθέσεις έχουμε ήδη ολοκληρώσει 17. Υπάρχουν και τέσσερις ε, τις οποίες ε, δεν ολοκληρώσαμε και γι' αυτό ακριβώς ε, δεν λάβαμε και την τελευταία δόση. αναγκαστήκαμε να λάβουμε κάποια επίγοντα μέτρα έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην... στην But it some spillover effect. τη ρευστότητα του προϋπολογισμού. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ε, όπου χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την δόση της μακροοικονομικής αρρωγής. Σας διαβεβαιώ όμως ότι εξακολουθούμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε και αυτά τα τέσσερα προαπαιτούμενα που δεν καταφέραμε να ολοκληρώσαμε, ολοκληρώσουμε και μάλιστα δύο από τα τέσσερα τα έχουμε ήδη ολοκληρώσει και τα άλλα δύο είναι πολύ κοντά. Ε, στην ολοκλήρωση. Η πρόθεσή μας ε, είναι να ολοκληρώσουμε όλα ε, τα προαπαιτούμενα από το προηγούμενο MFA έτσι ώστε να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα όταν θα εγκριθεί το καινούριο πρόγραμμα. Επίσης θα ήθελα να σας πω και δύο λόγια όσον αφορά το πρόγραμμα IMF διότι διασυνδέονται τα προγράμματα αυτά, όπως είναι και τα προγράμματα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ε, καθώς επίσης και άλλα διμερεί όργανα με τα οποία έχουμε σχέσεις. Ε, είμαστε πρόσφατα και στην ε, Ουάσιγκτον όπου συζητήσαμε και τις, τα προαπαιτούμενα για, το, για την επόμενη δόση και ευελπιστούμε ότι θα τα έχουμε ολοκληρώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόθεσή μας βεβαίως είναι και με την Ουάσιγκτον να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και περί τον Ιούνιο θα είμαστε σε θέση να ε, προχωρήσουμε ε, με την ε, επόμενη δόση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι ιδιαίτερος υποστηρικτικό, παρότι ένα από τα θέματα το οποίο είναι ιδιαίτερος βαρύ από πολιτική άποψη καλύπτει περίπου το 30%. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν όλες, να πάρουμε όλες τις δυνατότητες έτσι ώστε να μεταρρυθμιστεί το μέρος του φυσικού αερίου και ε, έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε αστάθεια ή οποιαδήποτε έλλειψη προμήθειας τούτων λεχθέντων. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας, αλλά να σας ζητήσω να μας υποστηρίξετε, να μας δώσετε τη στήριξή σας για μία ακόμα φορά ε, όσον αφορά την μακροοικονομική ε, αρρωγή MFA έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις αλλά και έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, ε, διασφαλίσουμε την ε, δημοσιονομική σταθερότητα της Ουκρανίας. ε, σας διαβεβαιώ ότι από τη δική μας πλευρά θα προσπαθήσουμε να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση έτσι ώστε την πρώτη δόση του MFA να την έχουμε όσο γίνεται ε, πιο γρήγορα και νομίζω ότι αυτό μπορεί να καταστεί δυνατόν στην αρχή του φθινοπόρου. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Ε, πολύ για την ενημέρωση. Εμείς δεν ασχολούμαστε με την εξωτερική πολιτική και δεν πειράζει να λέγω και πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, όχι γενικόλογα. Ε, θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα τέσσερα προαπαιτούμενα που δεν έχουν κλείσει και για ποιο λόγο δεν έχουν κλείσει και ποιε είναι οι επιφυλάξεις σας, για, να έχουμε πλήρη εικόνα και μετά θα πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. um... Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε για τέσσερα προαπαιτούμενα, δύο εκ των οποίων, να σας πω ποια είναι. Πρώτον, το θέμα της απαγόρευσης ξυλίας, το δεύτερο εκτιματολόγιο, συγγνώμη, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και αυτόματη ε, επαλήθευση ε, το πόθεν που ε, ε καταθέτουν ε, τα δημόσια πρόσωπα. Για να αποπολιτικοποιηθεί το θέμα αυτό, θα αναθεωρηθεί από ε, μια Επιτροπή Διατησίας αρμπιτράζ υπό τη Συμφωνία Σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιλέξαμε αυτό το δρόμο για να ε, βεβαιωθούμε ότι υπάρχει λύση. Αν είναι εντός της Συμφωνίας Σύνδεσης θα βρεθεί μια οριστική λύση και όχι ε, πολιτικοποιημένη. Ε, έγινε μια αλλαγή της νομοθεσίας, υιοθετήθηκε ένας νόμος στην αρχή του έτους ε, για την πιστοληπτική ικανότητα, ε, για το θέμα του τελικού δικαιούχου στις ιδιοκτησίες και όταν γίνεται λόγος για προαπαιτούμενα, θέλω να το τονίσω αυτό, αυτό το προαπαιτούμενο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο από την αρχή, δεν το είχαμε καταλάβει ε, με τον ίδιο τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες διαφορετικά. Τώρα τι σημαίνει η Ουκρανία. Δημιουργεί ένα νέο μηχανισμό που δεν υπάρχει πουθενά σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα δημιουργούμε προηγούμενο που θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Προφανώς χρειαζόμαστε βοήθεια ε, και εμπειρία για να μην είναι κακό το προηγούμενο. Έχουμε λοιπόν εμπειρογνώμονα δικό σας, ε, πριν από ένα μήνα ήρθε στην Ουκρανία και άρχισε να εργάζεται για το συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, αλλά τα προπετούμενα δεν μπορούν να ολοκληρωθούν όλα ταυτόχρονα και για την αυτόματη επαλήθευση των δηλώσεων πόθεν αλλάξαμε την προσέγγιση. Ασχολήθηκα προσωπικά ε, και ως αποτέλεσμα όλων αυτών όλα τα θέματα λύνονται. Έχουμε το πλαίσιο αναφοράς και η UNDP που είναι αρμόδια για ε, το λογισμικό προκήρυξε προχθές διαγωνισμό. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών δηλαδή. Ελπίζω να έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε τα προβλήματα, αλλά θέλαμε πιο συγκεκριμένες αναφορές. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο έχει η κυρία Ματάνοβα. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Χωρίς να μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες, θέλω να συμπληρώσω ότι πέραν από την ε, μακρονομική χρηματοδοτική στήριξη που πραγματικά έχει επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην οικονομία της χώρας, υποστηρίζουμε την Ουκρανία και με ένα μεγάλο ε, διμερές πρόγραμμα και εσείς άλλωστε πραγματοποιήσατε και μια επίσκεψη στην Ουκρανία πριν από ένα χρόνο και διαπιστώσατε και στην πράξη την ε, αρρωγή που παρέχουμε στη χώρα αυτή. Θέλω να πω ότι από το 2014, όταν ε, πραγματοποιήθηκε η επανάσταση του Μαϊντάν, υποστηρίζουμε ε, και ε, συμβάσεις οικοδόμηση κρατικών κτηρίων που επίση συνοδεύονταν από μια σειρά από προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα ε, ήμασταν πραγματικά πολύ χαρούμενοι <laughs> από πλευρά Κομισιόν για τις προϋποθέσεις που, που είχαν καταρτιστεί και πράγματι μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε οικοδομήσει ένα σημαντικό ε, σύνολο κτηριακών εγκαταστάσεων που ε, αφορούν την ε, αποκέντρωση, την καταπολέμηση της, ε, της διαφθοράς, δικαστήρια και αυτό βεβαίως συνδυάζεται και με το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο που έχουμε συνδιαμορφώσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης υπάρχει και μια μεταστροφή και κατευθύνουμε περισσότερη χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις και την οικονομική ανάπτυξη. Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουμε καταρτήσει και ένα σχετικό πρόγραμμα και πρόσφατα ε, καταρτήσαμε και ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή αποδοτικότητα που επίσης θα ενισχύσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Θέλω να υπογραμμίσω λοιπόν ότι σε όλα αυτά τα προγράμματα και όλα αυτά τα χρόνια ένα μεγάλο μέρος των πόρων κατευθύνεται προς τη συνεργασία με, και με τα κράτη-μέλη και με διεθνείς ε, ε οργανισμούς, ε, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Και όλα αυτά βεβαίως συμβαδίζουν και συνδυάζονται και με μεταρρυθμίσεις πολιτικής και με αντίστοιχα προαπαιτούμενα, όπου υποστηρίζουμε μια σειρά από κατευθύνσεις, στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με το Υπουργείο, ε, έχουμε καταρτήσει ένα ε, πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων δαπανών με τη συνεργασία της Σουηδίας, της Λιθουανίας, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μια σειρά από άλλους ε, κλάδους γίνονται αντίστοιχες κινήσεις Υπάρχει για παράδειγμα μεγάλη υποστήριξη από τη δική μας πλευρά προς την ενίσχυση των αρχών καταπολέμησης της διαφοράς. Συνεργαστήκαμε για το σκοπό αυτό με τις ε, κυβερνήσεις της Δανίας, της Πολωνίας και νομίζω και της Σουηδίας. Γενικά λοιπόν υπάρχει ένα... Ε, υπάρχει μια ολοκληρωμένη ένα ολοκληρωμένο σύνολο υποστηρικτικών προγραμμάτων που έχουμε καταρτήσει και αναπτύξει προκειμένου να ενισχύσουμε και να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ε, και εγώ κατάγομαι από χώρα της μετάβασης και πρέπει να πω ότι ε, το μέγεθος των μεταρρυθμίσεων που έχουν πραγματικά υλοποιηθεί, όχι στα χαρτιά, που έχουν υλοποιηθεί στην πράξη στην Ουκρανία, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πέρσι συνταξιδοτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ε, ε, μεταρρύθμιση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, πραγματικά μεγάλες μεταρρυθμίσεις ε, που ε, μάλιστα ακόμη και σε προηγμένες, ανεπτυγμένες χώρες θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνει κανείς τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις, τόσο βαθιές μεταρρυθμίσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια στην κυβέρνηση της Ουκρανίας. Γι' αυτό και εμείς Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με την χρηματοδοτική στήριξη που έχει υπάρξει από, την, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσει να συνεχίσει η χώρα. Αν ήταν απλό δεν θα ήμασταν εδώ εμείς. Αυτό είναι το θέμα. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη για τα τέσσερα ε, προαπαιτούμενα που είναι σε εκκρεμότητα και πότε υπολογίζεται να αποδεσμευτεί η δόση των 600 εκατομμυρίων. Ποια είναι τα εμπόδια ακόμα σε αυτό το δρόμο. Ε, ε, πρώτη ερώτηση. Και δεύτερη ερώτηση. Όλο αυτό το θέμα είναι πραγματικά πολύ επίπονο και πάντα επιπλήττονται αυτοί που δεν φταίνε. Αλλά στην επίσκεψή μας τι είδαμε. Υπάρχουν μεγάλες αντιστάσεις. Είχα μια συζήτηση με βουλευτές που μέχρι σήμερα δεν την έχω ξεχάσει ε, για την άρνηση, δημοσιοποίηση περιουσιακών στοιχείων κτλ. Και είχα την αίσθηση ότι όπου αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πόσο βιώσιμα θεωρείτε αυτά που έχουν επιτευχθεί. Και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο ότι δεν είναι απλώς στα χαρτιά, αλλά εφαρμόζεται. Αλλά με ποια βιωσιμότητα και ποια προοπτική γιατί μπορεί να υπάρξει και επιστοδρόμηση. Πώς το εκτιμάτε αυτό εσείς και εσείς κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Uh, how sustainable the... Πόσο βιώσιμες είναι οι μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το βλέπουμε κάθε μέρα, ότι στην Αμερική δεν έχει λυθεί αυτό. Είναι κάτι σχετικό η ε, βιωσιμότητα. Ε, υπάρχουν κάποιες μεταρρυθμίσεις που γίνονται για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά πολιορκούνται ε, σε πρώην πολύ δημοκρατικές κοινωνίες. Δεν μπορώ να προβλέψω τι μπορεί να συμβεί μετά από μια δεκαετία στην Ουκρανία. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι Και το υπενήχθη και ο Υπουργός όταν ε, αναφέρθηκε στο θέμα του πραγματικού δικαιούχου. Νομίζω ότι εμείς όταν ε, συγγράψαμε αυτά τα προαπαιτούμενα ήμασταν πάρα πολύ φιλόδοξοι γιατί στο προηγούμενο ε, πρόγραμμα μακροοικονομικής βοήθειας δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη, αυτό το προαπαιτούμενο. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να ελέγχει ποιο είναι ο τελικό δικαιούχο ενό περιουσιακού στοιχείου. Ούτε καν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν το κάνουν αυτό. Καμιά φορά νομίζω επιδεικνύουμε υπερβολικό ζήλο. Και καλό είναι να παραδεχθούμε ότι μπορεί να είχαμε επιδείξει και λιγότερη φιλοδοξία. Για το θέμα του πραγματικού δικαιούχου χαρτογραφήσαμε, ε, τα ύδατα Τώρα οι εμπειρογνώμονε συνεργάζονται με την κυβέρνηση για να βρεθεί ένας δρόμος που θα μα επιτρέψει να πούμε ότι έχει πληρωθεί το προαπαιτούμενο και να είναι όμως κάτι αξιόπιστο και σοβαρό. Στην περίπτωση επαλήθευση του πόθεν της τη δήλωση ε, περιουσιακών στοιχείων και πάλι είναι κάπως υπερβολικό και το εύρος και το βάθος το οποίο ψάχνουμε και ξεπερνάει τα όσα ισχύουν στη δική μου πατρίδα, δεν ξέρω στη δική σας ε, τι συμβαίνει. Είναι δύσκολη η υπόθεση και δαπανηρή και δύσκολη η υπαλήθευση. Άρα χρειάζεται ε, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αλλά διαπιστώνουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και δύσκολο να πληρωθούν αυτά τα Για Οι αντιστάσεις που αναφέρατε και είδατε κυρία Πρόεδρε, σε κάποιους θύλακες της Βουλής, τη Ράντα και σε κάποιους δημοσίους υπαλλήλους ή εξωματοχούς είναι ε, προφανής. Όταν έχεις μια χώρα σε μετάβαση, κάποια δρεωμένα συμφέροντα αντιστέκονται. Δεν θέλουν να υποχωρήσουν, να αποκαλύψουν τα περιουσιακά στοιχεία κτλ. Η συζήτηση γίνεται, είναι πάρα πολύ ζωντανή, πολύ έντονη και την υποστηρίζει μια πάρα πολύ ισχυρή κοινωνία των πολιτών στην Ουκρανία. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι σε ό,τι αφορά την αίσθηση ε, για την ύπαρξη της διαφθοράς είναι πάρα πολύ ψηλή αυτή στην Ουκρανία. Αλλά όσοι μελετούν συστηματικά τη διαφθορά γνωρίζουν ότι μόλις αρχίζει μια κυβέρνηση να καταπολεμάει τη διαφθορά εκτοξεύεται και η αίσθηση του κόσμου γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση δημόσια και κριτική και από εμά και από άλλους ζωρητές και βράζει κάπως εκεί η συζήτηση. το να δημοσιοποιούνται οι περιουσίες, το να είναι διαφανείς οι διαδικασίες βοηθάει πάρα πολύ. Ε, έχει υπάρξει μετατόπιση, ε, αλλαγή μοντέλου στην Ουκρανία. Κάτι που ήταν κρυφό και κάτω από το χαλί τώρα είναι τμήμα της δημόσιας συζήτησης και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης. Και τι γίνεται με τα υπόλοιπα τρία προαπαιτούμενα για τη μακροοικονομική βοήθεια. Α, για το παλαιό πρόγραμμα. Ε επιβεβαίωση, η του πόθεν υπάρχει. το μεγαλύτερο κομμάτι από το προαπαιτούμενο ήταν να δημοσιοποιείται αυτή η πληροφόρηση. Πριν από 1,5 χρόνο το έχουν κάνει και τώρα ε, προχωρούν ε, στην εκπόνηση αυτού του λογισμικού που ανέφερε ο υπουργό για να είναι αυτόματη αυτή η ε, ο έλεγχος του πόθεν έσχεση. Αντίστοιχο κάνει και το ελεγκτικό συνέδριο και για στην προετοιμασία τώρα για το νέο πρόγραμμα ακροοικονομικής βοήθειας επιμένουμε να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα αρχίσουν ε, ε τις σημαντικότερες υποθέσεις. Όχι με κάποιο διευθυντή σχολείου σε ε, ένα χωριό ή σε μια περιοχή που έχει 2.000 μαθητές. Από τα χοντράντος και τα πολιτικά να αρχίσουν και σε σχέση με ε, το λογισμικό νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Το δεύτερο για τον πραγματικό δικαιούχο ε, κάποιου περιουσιακού στοιχείου είναι πιο δύσκολο. Εκεί χρειάζεται τεχνική βοήθεια από πλευράς μας ε, που έχουμε παράσχει για να δούμε ποιες είναι οι δυσκολίες για να αρθούν και οι παρεθέσεις ας πούμε, που σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει και διαδικασία διατησίας υπό τη Συμφωνία Σύνδεσης και το Μητρό Δανείων επίσης έχει εγκριθεί. Credit Registry. Έχουν προχωρήσει λοιπόν και στα τέσσερα προαπαιτούμενα και θα πληρωθούν νομίζω όλες οι προϋποθέσεις. Τρία είναι τα μέλη της Επιτροπής μας που έχουν ζητήσει το λόγο συνάδελφος Τσέλερ που ήταν μαζί μας άλλωστε και στην Ουκρανία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ και σα ευχαριστώ που βρίσκεστε στη διάθεσή μας. Οι μακροοικονομικές και ε, ε, βοήθειες δίνονται προκειμένου να ε, στηριχθεί εν γέννη μια χώρα ε, και από άποψη χρηματοδοτική, χρηματοπιστωτική. Ο πληθωρισμό στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ ψηλό. Νομίζω ότι εξακολουθεί να κινείται στα επίπεδα του 14-15% και αυτό ένας από τους λόγους ε, που, που συνετέλεσε αυτό ήταν ε, και η ανεξέλεγκτη εκροή κεφαλαίων από την Ουκρανία. Υπήρξαν ε, χρεοκοπίες τραπεζών και στη συνέχεια τα περιουσιακά του στοιχεία βρίσκονταν κάπου στο εξωτερικό η διευθύντρια της Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Ρενιάτοβα, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, Ρενιάτιεβα, η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, είχε, έκανε κάποιες ε, ε, βελτιώσεις. Πώς προχωράει η διαδικασία αυτή, γιατί ξέρω ότι ε, πολλές ε, ρωσικές τράπεζες αλλά και αυστριακές τράπεζες έχουν παρουσία στην Ουκρανία πώς θα αποφευχθεί ε, στο μέλλον ε, η εκροή κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων από την Ουκρανία στο εξωτερικό. Κύριε Βόν, ευχαριστώ. Συμμετείχα και εγώ στην επίσκεψη αυτή και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πραγματικά διαπιστώσαμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Τα δύο πράγματα που με εντυπωσίαζαν ήταν πρώτον οι κατηγορίες για τη διαφθορά. Ε, σχημάτισα την εικόνα στο χρο... Ε, την στιγμή της επίσκεψης τουλάχιστον ότι πράγματι δεν έχει η χώρα την δυνατότητα αντιμετώπισης του μεγέθου του, του προβλήματος. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, σε, καμία περίπτωση δεν μπορούσαν μόνε τους να ε, αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δεύτερο θέμα είναι ότι τα, τα χρήματα του MFA πηγαίνουν στο κεντρικό προπολογισμό και γι' αυτόν τον λόγο μας υπόθηκε ότι ήταν πολύ δύσκολο να ειχνηλατηθούν τα, τα κεφάλαια αυτά, τα κονδύλια αυτά, να διαπιστώσει κανείς πού ακριβώς καταλήγουν. Ε, και όπως είπα λοιπόν, ακριβώς λόγω αυτού του προβλήματος θα με ενδιέφερε να μάθω αν έχουν γίνει ε, βήματα προόδου προκειμένου να ελέγχονται καλύτερα ε, το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα που ε, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την θέση της ε, Επιτροπής ε, όσον αφορά τα πρότυπα τα οποία είναι πολύ υψηλά, όσον αφορά τον ε, τελικό δικαιούχο. Και να σας εξηγήσω γιατί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια ειδική επιτροπή για θέματα φορολογικά. Και έχουμε και έναν κατάλογο ε, φορολογικών ε, παραδείσων ε, τον οποίο που παρακολουθούμε προσεκτικά, γιατί θέλουμε να δούμε πώς ακριβώς εργάζονται. Και επίσης είναι πολύ συγκεκριμένα τα κριτήρια έτσι ώστε να συμπεριληφθεί μια χώρα στους ε, φορολογικούς παραδείσους ε, και στη διάρκεια της εξέτασης ε, των Panama Papers είχαμε μελετήσει πάρα πολύ τα θέματα αυτά ε, και ε, διαπιστώσαμε ότι πολλοί, ε, πολλά υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη της Ουκρανίας είχαν ανοίξει, είχαν δημιουργήσει εταιρείε στον Παναμά που είναι σαφώς φορολογικός παράδεισος ακόμα και στη διάρκεια του πολέμου. Γινότανε πόλεμος και οι πολιτικοί δημιουργούσαν εταιρείε σε φορολογικό παράδεισο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση αυτή. Και επομένως είναι πολύ σωστό να υπάρχει αυτή ε, αυτό το προαπαιτούμενο. Ε, εάν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει χρήματα, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να λυθούν τα ζητήματα αυτά. Εδώ δεν υπάρχει υποψία διαφθοράς, υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία. Τα συζητήσαμε μάλιστα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι το θέμα του τελικού δικαιούχου, πραγματικού δικαιούχου, beneficiary owner, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, που είναι ένα σώμα που θέλει πραγματικά να καταπολεμήσει την διαφθορά. Από τεχνικής απόψεως, ε, λοιπόν, τα πρότυπα δεν είναι πολύ υψηλά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι έτσι ώστε να αναγνωρίσει κανείς τον τελικό δικαιούχο Βεβαίως ε, υπάρχουν προβλήματα παντού ε, όσον αφορά τον ε, τελικό δικαιούχο, αλλά τα προβλήματα δεν είναι τεχνικής φύσεως, είναι πολιτικής. Ναι, είναι πραγματικά σημαντικό να γνωρίζουμε και τους σιωπηρούς συμμετέχοντες για να αποφεύγονται και συγκρούσεις συμφερόντων. Είναι πραγματικά μία ε, από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις. Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και στο παρελθόν αρκετές φορές. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ε, περίμενα την επίσκεψή σας. Δεν ήξερα ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Πρέπει να το δω αυτό με το επιτελείο μου. Ήθελα να, να σας δω και στην Ουκρανία γιατί στο πλαίσιο αυτό έχουμε Ε, γιατί, ε, την, γιατί έχουμε τη δυνατότητα όταν βρισκόμαστε ε, κατά πρόσωπο να σας δείχνουμε και περισσότερα στοιχεία και να μπαίνουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Εν πάση περιπτώσει την επόμενη ε, επίσκεψή σας. Για την εκροή κεφλα, κεφαλαίων και πώς θα εξασφαλίσουμε να εμποδιστεί η ανεξέλεγκτη εκροή κεφαλαίων από τη χώρα. Καθώς και ε, πού βρισκόμαστε στην μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος. Πραγματικά, η προηγούμενη διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας απέδειξε μεγάλη ε, γενναιότητα, θάρρος, επέφερε πολύ σημαντικές αλλαγές, αντιμετώπισε χρονίζοντα προβλήματα και επετέφθηκαν πολλά πράγματα. 90 τράπεζες αφαιρέθηκαν από το τραπεζικό σύστημα. Μαζί λοιπόν προχωρήσαμε και στην εθνικοποίηση της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που κάναμε μαζί. Αυτά τώρα έχουν ολοκληρωθεί. Το τραπεζικό σύστημα είναι καθαρό πια. Η μεγαλύτερη ε, τράπεζα που βρισκόταν υπό την ιδιοκτησία δύο ολιγαρχών, πλέον τελεί υποκρατική ιδιοκτησία και ελέγχουμε το 55% συνολικά ολόκληρου τραπεζικού συστήματος από την κυβέρνηση. Άρα, το ερώτημα που θέσατε απευθύνεται στην πραγματικότητα με δύο τρόπους και σε εμάς ακριβώς γιατί είμαστε και εμείς μέτοχοι στο 55% των ε, τραπεζών αυτών. Πρόσφατα λοιπόν έχουμε εγκρίνει μια στρατηγική που θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα και που θα καταλήξει στην ε, διαμόρφωση και το μετασχηματισμό τολμώ να πω, ολόκληρου τραπεζικού συστήματος με διαφάνεια θα προχωρήσουμε στην επανειδιωτικοποίηση των κρατικοποιημένων τραπεζών και ελπίζουμε και οι ευρωπαϊκές τράπεζες να δείξουν ενδιαφέρον. Αυτά ως το τραπεζικό τομέα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα προβλήματα που ε, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν για να εμποδιστεί η εκροή κεφαλαίων για παράδειγμα τα BAPS. Επίσης, ε, έχουμε συνάψει μια σειρά από συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης, ακολουθούμε τις προδιαγραφές του ΟΣΑ, γιατί ξέρετε τα, στις εκροές ε, κεφαλαίων τα χρήματα δεν πηγαίνουν, πρώτα, ε, δεν πηγαίνουν κατευθείαν στις offshore, πηγαίνουν πρώτα σε χώρες όπου υπάρχουν ε, χαμηλότερες, χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές. Άρα έχουμε έρθει και σε συμφωνία με χώρες όπως κάτω χώρες, η Κύπρος και καταρτήσαμε και έναν νόμο ο οποίος απαντά σε όλα αυτά τα θέματα. Ε, έχει τη μορφή νομοσχεδίου αυτή τη στιγμή, έχει υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να εγκριθεί σύντομα. Αυτά για τις εκλογές κεφαλαίων. Για τη διαφθορά τώρα. Μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα από αυτά που ακούστηκαν ήδη. Έχω και προσωπική εμπειρία από αυτό το θέμα. Προτού γίνω υπουργό. Ε, εγώ ήμουν ε, αξιωματούχος της κρατικής διοίκησης, δούλευα στην Κρέκα ε, και συνέβαλα στην δημιουργία της αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς. Η αρχή καταπολέμησης του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, για παράδειγμα, ήταν σημαντικό βήμα. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εξαρτήσεις και διασυνδέσεις. Όταν λέμε λοιπόν ότι ε, είναι απαραίτητο να καταπολεμηθεί η διαφθορά, δεν είναι απλά λόγια αυτά. Προβαίνουμε στην πράξη και τα κάνουμε αυτά. Γιατί βλέπουμε ένας οργανισμός, για παράδειγμα, να εντοπίζει περιπτώσεις διαφθοράς. Ε, υπάρχουν και οι άλλες εθνικές αρχές αλλά το σημαντικό, το σημαντικότερο στοιχείο από τη δική μας ε, σκοπιά είναι η θέσπιση του ειδικού δικαστηρίου για την, ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί αυτό ήταν και ένα αίτημα της επανάστασης του Μαϊντάν, αν θέλετε. Ήταν βεβαίως και η ευρωπαϊκή η ευρωπαϊκή προοπτική της, ε, της Ουκρανίας, αλλά ήταν και όχι απλά η δυσαρέσκεια, αλλά η οργή για την έκταση της διαφθοράς στη χώρα. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε όλα αυτά τα βήματα και νομίζουμε ότι η δημιουργία, η ίδρυση αυτού του ειδικού δικαστηρίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι σοβαρή, σοβαρό βήμα προς την κατεύθυνση που έχουμε χαράξει. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να καταπολεμηθεί επιτέλους μέχρι τέλους η διαφορά στη χώρα. Άρα, η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι ένα πραγματικό θέμα που μας έχει απασχολήσει. Η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης Διαφοράς δημιουργήθηκε τώρα, πρόσφατα. 600 ανθρώπους εκπαιδεύσαμε, ήταν νέοι όλοι τους, Καταρτίστηκαν όμως, εκπαιδεύτηκαν και πλέον έχουν διασπαρεί σε όλες τις εθνικές αρχές και σε όλα τα θεσμικά όργανα της χώρας μας προκειμένου να βοηθούν και να παρακολουθούν και να ελέγχουν την καταπολέμηση διαφθοράς. Διαφάνεια και εκτέλεση προϋπολογισμού, ιδίως όσον αφορά τη διάσταση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής στήριξης. Εγώ ως υπουργό, ελπίζω να με καταλαβαίνετε, είμαι υποχρεωμένος να εξασφαλίζω ότι όλα τα χρήματα που έχουμε στον προϋπολογισμό αξιοποιούνται. Βεβαίω με έλεγχο του πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα στη βάση προτεραιοτήτων και να ελέγχουμε και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτό το μηχανισμό στι χώρε. Γιατί προφανώ δεν μπορούμε να ιχνηλατούμε ούτε να παρακολουθούμε όλα τα χρήματα που έρχονται στον προπολογισμό. Πρέπει να υπάρχει και κάποια εμπιστοσύνη και από τη δική μα πλευρά και από τη δική σα πλευρά για το πώ εισραίουν και πώ δαπανώνται τελικά τα χρήματα του προπολογισμού. Υπάρχουν αρχέ. Υπάρχει για παράδειγμα η Γενική Εισαγγελία που βεβαίω πρέπει να ε, μεταρρυθμιστεί πλήρω. Έως τότε ε, περιορίζω εγώ, σα το λέω καθαρά, κάποιε επενδύσει που θα μπορούσαν να γίνονται ακριβώ γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα γίνουν σωστά οι επενδύσει αυτέ με καταπολέμηση της διαφθοράς. Άρα, το MFA πηγαίνει στον, στον προπολογισμό. Δεν ξέρω πώ ακριβώ θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ειχνηλασιμότητα, αλλά πρέπει να καταλάβετε πώ πώς, διαχειρίζεται μια χώρα τα χρήματά τη. Για τα Panama Papers. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχετε δίκιο. Πρώτον, σχετικά με το γεγονό ότι όταν αποκαλύπτονται κάποιε πληροφορίε πρέπει να υπάρχει αντίδραση, ε, μπορώ να σα πω ότι ε, δεν υπάρχει μόνο ένα τρόπο αντίδραση. Και νομίζω ότι ένα από τα βασικά στοιχεία τη επόμενη περίοδου είναι οι επερχόμενε εκλογέ. Αν δεν είναι σημαντικό αυτό για του Ουκρανού και δεν φανεί κάτι τέτοιο στι εκλογέ, γιατί να είναι σημαντικό για, για, όλο, για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αποκαλύφθηκαν κάποιε πληροφορίε, έχουν γνωστοποιηθεί. Ο Ουκρανικό λαό θα κρίνει πλέον. Του χρόνου θα γίνουν εκλογέ. Υπάρχει πολιτική βούληση. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει πολιτική βούληση να καθαρίσουμε το σύστημα να εξασφαλίσουμε ότι θα καταβάλλονται οι φόροι, ότι τα χρήματα θα μένουν στη χώρα. Υπάρχει αντίσταση. Ναι, τεράστια μάλιστα. Αλλά βήμα προς βήμα σημειώνουμε πρόοδο, προχωράμε και ο Ουκρανικός λαός θα κρίνει αν πετύχαμε τους στόχους μας ή όχι. Για τα τεχνικά θέματα μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ακόμη τεχνικές δυσκολίες. Είναι πολύ δύσκολο ε, ειδικά όταν υπάρχει αλυσιδωτή ιδιοκτησία, να αποδείξει κανείς ότι κάποιο συγκεκριμένο άτομο, άτομο είναι ιδιοκτήτη ενό περιοριστικού στοιχείου. Διότι αν έχει διαρρεύσει ένα όνομα μέσα των Panama Papers ως ιδιοκτήτη ε, μιας επιχείρησης ενός περιο... ή ενός περιουσιακού στοιχείου, αυτό είναι ένα στοιχείο. Αλλά προφανώς από την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών, πολλοί έχουν προβεί στην δική τους ανάλυση της πραγματικότητας και αποφεύγουν πλέον να δημοσιοποιούν τέτοιες ε, πληροφορίε. Άρα το πρόβλημα του εντοπισμού του πραγματικού κατόχου ή διοκτήτη ενός περιουσιακού στοιχείου έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο. Πώς θα το λύσουμε? Μαζί πρέπει να το κάνουμε, συνεργασία. Και πρέπει νομίζω να αποδεχθούμε ότι θα είναι μια διαδικασία που θα βρίσκεται διαρκώς υπό εξέλιξη. Δεν μπορεί να, να θεωρούμε ότι θα βρούμε μία λύση και θα τελειώσουμε. Και είναι και παγκόσμιο το πρόβλημα. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Υπουργέ, σα ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα. Α αρχίσω από την ερώτηση του κύριου που χρειάστηκε να φύγει για τη μακροοικονομική βοήθεια είναι ένα εργαλείο αντιμετώπιση των δυσκολιών ε, ισοζυγίου πληρωμών και φυσικά τον προπολογισμό αφορά γιατί ο προπολογισμό έρχεται να καλύψει τα προβλήματα ε, στις πληρωμές και η Ουκρανία είναι πολύ ψηλά στις χώρες στη διαφάνεια του προϋπολογισμού παγκοσμίω και δύο στοιχεία ανέφερε ε, το ένα ο Υπουργός είναι τα εξής, το δεύτερο το ανέφερε την τελευταία τριετία Ε, όντας σε πόλεμο μειώθηκε σε 1,7% το έλλειμμα του υπεροπλογισμού από 10 και παραπάνω. Ε, υπερπενταπλάσια είναι η μείωση, ε, δηλαδή και είχαν και πόλεμο και το 5% του ΕΠ πήγαινε σε πολεμικές στρατιωτικές δαπάνες. Καταλαβαίνουμε από τα στοιχεία τι σημαίνει αυτό για τις εξελίξεις στη χώρα, αλλά ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι την τελευταία τριετία οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν κατά 13% ε, από 53% έχουν φτάσει στο 40%. Είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά τα στοιχεία περί στολή των δημοσίων δαπανών. Όσοι από εμά παρακολουθούμε τις ηρωικές προσπάθειες του Γάλλου Προέδρου να ε, περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες κατά 1 ή 2% που έχουν τις υψηλότερες δημοσίες δαπάνες στη Γαλλία και βλέπουμε ποια είναι η αντίδραση του λαού, καταλαβαίνετε τι σημαίνει μέσα σε τρία χρόνια περιορισμός των δημοσίων δαπανών κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες. Βεβαίως εμείς το γενικό προϋπολογισμό υποστηρίζουμε γιατί από εκεί καλύπτονται οι ε, ε στο ισοζύγιο πληρωμών. Αλλά στα πλαίσια της διαφάνεια του προπολογισμού η Ουκρανία είναι από τους... Ε, καλύτερους ε, μαθητές ε, στα όσα παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ε, ιστορικά, όταν είναι ισχυροί οι θεσμοί σε μία χώρα, Τι χρειάζεται να έχουν διοκτικές αρχές πολύ καλές ερευνητικές και επιβολής του νόμου και να πατάσετε η διαφθορά τη στιγμή που ε, συντελείται. Ε, προχωράει αυτό στην Ουκρανία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Μόλις τώρα έγιναν οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, ε, θα πρέπει να συσταθεί δικαστήριο κατά της διαφθοράς. Εμείς είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό και ευθυγραμμιζόμαστε και με τη διεθνή κοινότητα, το διεθνές νομισματικό ταμείο ε, έχουν το ερευνητικό σώμα ε, για την διαφθορά, αλλά κάπου στη συνέχεια στη δικαιοσύνη χάνεται αυτό, διαχέεται. Η Ουκρανία ήταν πάρα πολύ επιτυχής μέχρι στιγμής στο εξή. Περιόρισε τις δυνατότητες, ε, τις ευκαιρίες διαφθοράς και το γεγονός ότι μειώθηκαν οι δημόσιες δαπάνες από το 53% στο 40% του προϋπολογισμού δεν σημαίνει μόνο οικονομίες και σημάζεμα του προϋπολογισμού, αλλά ότι κλείσανε και τις πόρτες της διαφθοράς. Πού υπήρχε περισσότερη ε, διαφθορά και που έγινε η διατησία. Στην ισοτιμία ε, του ε, νομίσματος ε, που ήταν σταθερή για να μην υπάρχουν κερδοσκοπίες. Το δεύτερο είναι ο τραπεζικός τομέας, το είπε ο Υπουργός. Αφαιρέθηκαν πάνω από 90 ε, άδειε τραπεζών. Η προληπτική εποπτεία ε, είναι πάρα πολύ αυστηρή, δρακόντη. Και το πρόβλημα είναι ε, ότι δεν υπάρχει ρευστότητα προς την πραγματική οικονομία γιατί είναι πολύ υψηλέ οι απαιτήσει για τις εγγυήσεις κτλ. Και έχουν ε, ε, πλεόνασμα στη ρευστότητα οι τράπεζες, δεν έχουν πρόβλημα. Άρα πατάχθηκε η διαφθορά στις τράπεζες. Ο τρίτος τομέας ήταν κάτι για το οποίο επιβραβεύτηκαν διεθνώς εισαγωγή ηλεκτρονικών ε, ε, διαγωνισμών. Ε, προς όλο λέγεται αυτό το σύστημα. Περίπου 1% το έπιν, οι οικονομίες που έγιναν από τις δημόσιες συμβάσεις χάρη στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, προκηρύξεις κλπ. Θα ενταχθούν και άλλα στοιχεία στο σύστημα. Επιστροφές ΦΠΑ, άλλος θύλακος διαφθοράς. Και αυτό θα γίνει αυτόματα πλέον έτσι ώστε να ε, παταχθεί η διαφθορά και να εξαφανιστεί. Τώρα σε ποσοστό του ΕΠ δεν ξέρω, να σας δώσω άλλο στοιχείο. Ελήφθη μια απόφαση από την κυβέρνηση Γκρόισμαν ε, το Μάιο του 2016 να εξισώσει το τιμολόγιο φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά με το βιομηχανικό τιμολόγιο. Ε, αυτό σημαίνει ότι τελείωσε η διαφθορά μέσα σε μία μέρα, από τη μία μέρα στην άλλη. Η Ναυτογκάζ, το μονοπόλιο του φυσικού αερίου, είχε απώλειες 18 δισεκατομμύρια το ένα έτος και το επόμενο ένα, ένα δισεκατομμύριο κέρδη. Δημιουργείται έτσι μια πυραμίδα στη γραφική παράσταση, ένα δέλτα, ε, που δείχνει πώς ε, ε, καταπολεμήθηκε η διαφθορά και πώς οδηγήθηκε η ναύτογκα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή χρειάζονται θεσμοί που θα υποστηρίξουν και την καταστολή και το σκέλος της επιβολής κυρώσεων. Κάποιος κύριος από την Πορτογαλία ερώτησε κάτι. Υπάρχει σήμερα στην Ουκρανία διαφθορά βεβαίως. Υπάρχουν ισχυροί ολιγάρχε, βεβαιότατα. Εγώ θα πρόσθετα ότι είναι αρκετά φτωχότεροι από ό,τι πριν από τρία χρόνια, αλλά είναι βαθύπλουτοι έτσι κι αλλιώς. Ε, στα έγγραφα του Παναμά μπορεί να είδατε, θα έχετε σίγουρα δει και ουκρανικά ονόματα. Αλλά όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοστατεί στην προσπάθεια αυτή ε, γιατί το θέμα των μη συνεργαζομένων κρατών ε, σε θέματα καταπολέμησης ε, της διαφθοράς και στις χώρες ΝΙΕ υπήρχαν χώρες που ήταν πρώτα στη μαύρη λίστα, τώρα στην κρίζα. Δεν είναι Ουκρανία μία από αυτές, ως χώρα, ναι. Αλλά ε, βεβαίως υπάρχουν ε, μεμονωμένα άτομα που έχουν κρυφά περιουσιακά στοιχεία και ε, κρυμμένα και βαθύπλουτα σε φορολογικούς ε, παραδείσους, αλλά ως χώρα η Ουκρανία δεν συζητήθηκε ποτέ να ενταχθεί στον κατάλογο των χωρών που δεν συνεργάζονται για τη φοροδιαφυγή. Και, όπως σας είπα, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μεγάλη προτεραιότητα και μεγάλη εμβληματική μάλιστα προτεραιότητα. Με την κυβέρνηση της Δανίας συνεργαζόμαστε για να τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν τους θεσμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε ε, που ήρθατε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση και την ανταλλαγή. Θα παραμείνουμε σε επαφή. Είδατε ότι δουλειά έχουμε. βεβαίω θέλουμε να σα αθαρρύνουμε, να συνεχίσετε σε αυτό το δρόμο. Πολλοί μα έχουν εντυπωσιάσει αυτά που ακούμε. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά που έχετε. Αν λέτε και ο ίδιο ότι έχετε επιτύχει κάποια πράγματα, είμαστε κι εμεί ικανοποιημένοι. Θα σα συνοδεύσουμε σε αυτή την πορεία και με τη μελέτη που θα γίνει περί τα τέλη του έτου. Ευχαριστώ πολύ που μα ήρθατε. Καλή σα επιτυχία και στο καλό. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης, το σημείο 7, ειδική έκθεση 7 του 2018 για την ε, Τουρκία. Η κυρία Γιάκοψεν έχει αναλάβει την παρουσίαση. Πολύ σύντομα, κανείς άλλος δεν θα πάρει το λόγο εκτός από, την, ε, από το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου, την κυρία Γιάκοψεν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτή την ειδική έκθεση για την προεντεξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία, το IPA. Η δημοκρατία της Τουρκίας παραδοσιακά διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις, είναι βασικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην άμυνα, στο εμπόριο και από το 1999 αποτελεί υποψήφια προσένταξη χώρα. Σε συνεργασία λοιπόν με τις τουρκικές αρχές, η πρωτεξιακή βοήθεια αποτελείται από προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Κομισιόν σε μια μεγάλη πλειάδα τομέων πολιτικής, όπως είναι το κράτος δικαίου, η διακυβέρνηση, η γεωργία, οι υποδομές και ε, η ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Η Τουρκία είναι ο πρώτος δικαιούχος ε, ευρωπαϊκής βοήθειας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 7-13 η, τα κονδύλια προς την Τουρκία ανήλθαν σε 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ και για το ε, επόμενο διάστημα 14-20 ανήλθαν στα 4,5 δισεκατομμύρια. Η πρόοδος ε, στις προενταξιακές δραγματεύσεις είναι πάρα πολύ αργή και ε, έως το 2015 είχαν ανοίξει μόνο 16 από τις 35 κεφάλαια και μόνο ένα έχει κλείσει. Από τον Ιούλιο του 2016 και, την, και το πραξικόπημα που έγινε στην Τουρκία, η Τουρκία έχει εισέλθει σε μια κατάσταση έκτακτης ε, ε, ε ανάγκης και έκτακτης κατάστασης και αυτό οδήγησε στην αναστολή ευρωπαϊκής ε, βοήθειας. Κάτι που το εξετάσαμε στη διάρκεια της, του ελέγχου μας. Στόχος μας ήταν ε, να ε, διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα της προληπτικής βοήθειας, σκοπός της οποίας είναι να βοηθήσει τη χώρα να συγκλίνει με το κεκτημένο και να ενισχύσει τις διοικητικές της ικανότητες. Εξετάσαμε αν το IPA είχε το σωστό σχεδιασμό και αν η προληπτική βοήθεια ήταν αποτελεσματική ως προς το στόχο της να υποστηριχθούν οι προτεραιότητές της στην Τουρκία. Ποια είναι τα πορίσματά μας λοιπόν. Συμπεραίνουμε ότι οι στόχοι IPA είχαν σχεδιαστεί επαρκώς και ορθώς από την Κομισιόν. Ωστόσο, τα πρωτεξιακά κονδύλια που δαπανήθηκαν στην Τουρκία δεν κατάφεραν να ε, ανταποκριθούν σε κάποιες βασικές αρχές όπως είναι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την ενίσχυση της ε, κοινωνίας των πολιτών. Τομείς όπου ε, είναι αναγκαίοι και υπερόριμοι ε, υπερόριμες αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Βλέπουμε ότι η Τουρκία ή μάλλον η Κομισιόν δεν έχει εφαρμόσει επαρκώς τα κριτήρια που είχαν καταρτιστεί στους τομείς όπου δεν ήταν επαρκής και ικανοποιητική η πρόοδος. Η Κομισιόν λοιπόν πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση κονδυλαίων από τις εθνικές αρχές ή να προβαίνει σε διορθωτικά μέτρα όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η δυνατότητα αναστολής χρηματοδότησης όταν δεν πληρούνται οι αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν αντικατοπτρίζονται ρητός στον κανονισμό IPA. Όσον αφορά την εφαρμογή ε, οι έλεγχοι ε, ε, κατέληξαν στο ότι τα αποτελέσματα που επιδιώκονταν γενικά είχαν επιτευχθεί. Στα 13 από τα 14 υποεξέλιξη προγράμματα που ελέγξαμε, οι Κομισιόν και οι τουρκικές αρχές είχαν καταφέρει να καταρτήσουν σχέδιο για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, αλλά 8 από αυτά παρουσίαζαν καθυστερήσεις. Διαπιστώσαμε λοιπόν σημαντικές καθυστερήσεις ιδίω λόγω έλλειψη πολιτική βούληση των τουρκικών αρχών και λόγω βεβαίω και των πρόσφατων εξελίξεων στη χώρα. Τέλο, ε, τίθεται σε κίνδυνο και η βιωσιμότητα αυτών των προγραμμάτων λόγω της οπισθοδρόμησης που ε, διαπιστώνεται στις μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά λοιπόν την προενταξιακή πορεία της Τουρκίας, καταλήξαμε σε πέντε συστάσεις προς την Κομισιόν. Το IPA θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τομείς όπου οι μεταρρυθμίσεις είναι υπερόριμες, η Κομισιόν πρέπει να βελτιώσει, να βελτιώσει την τομεακή της προσέγγιση προκειμένου να επιτύχει τα βασικά χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν. Η Κομισιόν πρέπει να ενισχύσει την ε, χρήση πολιτικών ε, ε, προϋποθέσεων, να βελτιωθεί η παρακολούθηση και να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις μέσω της άμεσης διαχείρισης των κονδυλίων που έχουν χορηγηθεί. Η Κομισιόν απεδέχθη όλες τις συστάσεις μας και θέλω να την ευχαριστήσω για την επικοδομητική της στάση σε όλη τη διάρκεια αυτού του ελέγχου. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και αν έχουμε χρόνο είμαι στη διάθεσή σας και για ερωτήσεις που ενδεχομένως έχετε από αυτής της έκθεση. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο την Κλάουδια Σμιτ που είναι η συγκήτρια για το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι είναι μια σύντομη παρουσίαση της ειδική έκθεσης. Παρακαλώ, Κλάουδια Σμιτ. Σύντομα. Σύντομη παρουσίαση με πάρα πολλές παρατηρήσεις όμως ε, και αστερίσκους δυστυχώς. Ε, οι εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου πάντα είναι για μένα πολύ ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές. Η συγκεκριμένη με απογοήτευσε πάρα πολύ. Γιατί σε αντίθεση με τα όσα μόλις μας είπε το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, εγώ δεν τη βλέπω και τόσο θετική την έκθεση αυτή. Ούτε σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ούτε σε ό,τι αφορά τις δράσεις, για να μην πω την αδράνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, πραγματικά προκαλεί φρίκι να διαβάζουμε ε, έτσι ρητά αυτά που υποθέταμε, αλλά τα έχει διαπιστώσει, τα έχει αποκαλύψει το ελεκτικό συνέδριο. Ε, συνοπτικά. Θέλω να σας παραθέσω κάτι. Στην πραγματικότητα, στη χρήση των κονδυλίων στους στόχους είπα ένα, δεν ελήφθη υπόψη καθόλου ένα προαπαιτούμενο που είναι η ανεξαρτησία και μεροληψία της δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο και του οργανωμένου εγκλήματος, η ελευθεροτυπία, η ε, αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, η ενίσχυση των εξωτερικών ελέγχων και της κοινωνίας των πολιτών. Σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόοδη σε αυτό το τομέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ανεπαρκής οι τουρκικές αρχές δεν έχουν την πολιτική βούληση για να τελοποιήσουν όλα αυτά. Και μόνο λοιπόν η πρόταση αυτή θα σήμαινε για μένα ότι ε, άμα δεν το θέλουν και αυτοί, να σταματήσουμε όλη τη φασαρία και το θέατρο και να τα μαζέψουμε. Είναι πάρα πολύ απογοητευτικό αυτό που διαβάζουμε για όλα τα έργα, εκτός από ένα, ότι λείπει πολιτική βούληση και για τα υπόλοιπα είναι πολύ λίγοι οι υπάλληλοι, διοικητικοί μηχανή και τέτοια. Αλλά εμείς δαπανάμε εδώ ποσά πέραν ε, το λογικό. Και η Τουρκία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο να τα υπερισπιστεί αυτά. Ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι και ο Αυστριακό Επίτροπο Ιωάννη Χαν που τα βλέπουν κάπω διαφορετικά τα πράγματα από μένα γιατί μπορεί να έχουν ακόμα την ελπίδα ότι έχει ενδεχομένω νόημα να συνεχίσουμε τις προενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αλλά πόσα χρόνια επιτέλους θα διαπραγματευόμαστε. Από το 99 κρατάει αυτή η ιστορία και επιδεινώνεται συνεχώς αντί να βελτιώνεται η κατάσταση. Ε, κάποια στιγμή δεν θα πρέπει απλώς να αναβληθεί η εκταμείευση των κονδυλίων να τερματιστεί. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους πρόσφυγες ή τους προσφυγικούς καταβλισμούς στην Τουρκία. Είναι τελείως ξεχωριστά τα θέματα, να τα κρατάμε αυστηρά ξεχωριστά. Εκεί μπορεί να υποστηρίζει ε, η Τουρκία ε, την Ευρώπη, αλλά όχι με προοπτική την ένταξη. Δεν έχω ακούσει πολλά πράγματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μου αρκεί αυτό που λένε και παραθέτουν στη συστάσεις το ελεγκτικό συνέδριο για το πώς θα δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, συμφωνεί με τις συστάσεις, συμφωνεί με τις συστάσεις. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, τι κάνει η Κομισιόν. Άμα συμφωνεί με τις συστάσεις αλλάζει τίποτα. Δεν έχω ιδέα τι κάνει. Ερωτώ λοιπόν, τι σημαίνει αυτό πάρα πολύ συγκεκριμένα. Αν συμφωνεί με τις συστάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνει γνώση. Επόμενο θέμα αυτά τα προαπαιτούμενα και η ερεσιμότητα του προενταξιακού μέσου είπα, Δεν αξιοποιείται καθόλου. Ιδιαίτερα όταν δεν είναι επαρκής η πρόοδη. Γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτή η αιρεσιμότητα. Γιατί δεν καταφεύγουμε σε αυτή η επανασυγκέντρωση όπως ονομάζεται. Υπάρχει στο ΙΠΑ 1 δυνατότητα αναβολής της χρηματοδότησης σε περίπτωση που δεν τηρούνται ε, οι αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Και στο ΙΠΑ 2, στον αντίστοιχο κανονισμό, δεν αναφέρεται ρητά αυτή η πρόνοια. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι είναι τεράστια η επιπολαιότητά μας για ε, τα ποσά για τα οποία πρόκειται και διαπραγματευόμαστε και διαπιστώνουμε ότι δεν σε θέλει ο εταίρος, βρε παιδάκι μου και μάλλον στρέφεται ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση και σου γυρνάει την πλάτη. Ε, τότε θα πρέπει να σταματήσουμε να ε, γελιόμαστε και να βαφκαλιζόμαστε. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Madam Chair. Κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μέσα από αυτήν την διαδικασία είχαμε εξαιρετική συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο και θα ήθελα να το υπογραμμίσω και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ε, και τους ε, συναδέλφους της γι' αυτό. Κυρία Σμιτ, Συμμεριζόμαστε αυτήν την αγωνία σας και τον προβληματισμό σας για την Τουρκία βάσει των νέων στοιχείων. Ε, νομίζω ότι εδώ μπορούμε ε, εύκολα να κάνουμε και τη σύγκριση με την προηγούμενη συζήτηση ε, που είχαμε για την Ουκρανία. Στη μία περίπτωση όλοι αγωνίζονται έτσι ώστε να προχωρήσουν. Στην Τουρκία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και έχουμε πολύ κακές επιδόσεις. Ε, και πρέπει να σας πω ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία συνεχίζουν την προσπάθεια ε, όσον αφορά ε, για τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσαμε συγκεκριμένα στις συστάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου να σας πω τα εξής. Ε, πρώτα απ' όλα, ήδη το 2017 μειώσαμε ε, την ε, χρηματοδότηση κατά 89 εκατομμύρια ευρώ και στο στρατηγικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Επίτροπος Χάν τον Μάρτιο, στις 20 Μαρτίου συγκεκριμένα ήταν εδώ και έκανε την πρόταση της Κομισιόν να μειώσει 759 εκατομμύρια ε, από το ε, ε, μέσο IPA έτσι ώστε να φτάσουμε στα 253 ανά έτος για το, από το 20 και μετά. Στην ουσία δηλαδή συμφώνησε και το, ήταν και η, θέση της κυρίας Σάκε ότι είναι απαραίτητο να ξαναδούμε το σύνολο του, της χρηματοδότησης ε, IPA ε, γιατί ε, εκεί στην Τουρκία λείπει η πολιτική βούληση. Είναι σαφές για μεταρρυθμίσεις, άρα πρέπει να μειωθεί η χρηματοδότηση. Δεύτερον, την ε, βοήθειά μας ε, την ε, προσανατολίσαμε προς τη δημοκρατία, την προστασία και την συμμετοχή, την προστασία των πολιτών της, και συμμετοχή της κοινίας των πολιτών κτλ. Δηλαδή την προσανατολίσαμε προς συγκεκριμένα ζητήματα και στο επόμενο MFF προτείνουμε την βοήθεια να την επικεντρώσουμε στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Κατά την έννοια αυτή σταματήσαμε ε, να χρηματοδοτούμε ένα πρόγραμμα ε, στο δικαστικό τομέα ακριβώς λόγω της επιστοχώρησης που διαπιστώσαμε στον τομέα αυτό και ακριβώς λόγω των προβλημάτων ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης ε, και την κατάσταση με τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Επίσης εστιάσαμε περισσότερο στα προαπαιτούμενα όσον αφορά την προσέγγιση μας και όλο και περισσότερη προσοχή θα δίνουμε ακριβώς σε αυτήν την διαδικασία αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε πάρει ήδη κάποια βήματα έτσι ώστε να αυξήσουμε το ποσοστό ε, των χρημάτων ε, που ε, υπάρχει, για τα οποία υπάρχει έμεση διαχείριση από τις διαχειριστικές αρχές ενώ μειώσαμε τα χρήματα τα οποία η τουρκική κυβέρνηση άμεσα διαχειρίζεται. Ε, ε επίσης ε, πολλά στοιχεία τα ξαναφέραμε ε, στην Κομισιόν και στην διαχείριση δηλαδή της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χώρα αυτή γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει όλο και λιγότερη άμεση διαχείριση να έχει η Τουρκία. Ευχαριστώ. Ε, τελείωσε εδώ το θέμα στην ημερησία διάταξη. Σύντομη παρουσίαση σημαίνει αυτό, σύντομη παρουσίαση. Αλλά θα το γράψουμε ξανά στην ημερησία διάταξη γιατί πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Τι κάνουμε με όλο αυτό το ζήτημα. Και... Ζητώ συγγνώμη, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα να δώσουμε το λόγο στα μέλη. Αλλιώ θα παραταθεί η συζήτηση ε, Μόνο 15 λεπτά είναι σύντομη παρουσίαση, ακούμε τις παρουσιάσεις και δεν μπαίνει κανένα άλλο στο λόγο. Ολοκληρώνεται λοιπόν το θέμα αυτό τη ημερήσιας διάταξη και η δημόσια ε, συνεδρίαση. Παρακαλώ να αποχωρήσετε όλοι εκτός από τα μέλη τη Επιτροπή και εκείνοι που δικαιούνται να παραμείνουν. Και φυσικά οι σύμβουλοι. Και όλοι οι υπόλοιποι στο καλό. Ευχαριστώ και αν γίνεται αθόρυβα. Παρακαλώ να σταματήσει και η μετάδοση στο διαδίκτυο. Για να αρχίσει η κυκλισμένα των θυρών συνεδρίαση.